Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ, καθίστε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Καλωσορίζομαι θερμότατα τη Ρουμανική Προεδρία. Είναι η πρώτη συνεδρίαση της ΣΥΤΡΕ παρουσία εκπροσώπων της Ρουμανικής Κυβερνήσεως. Χαιρόμαστε όλους ιδιαίτερος που σας έχουμε εδώ. Για μας είναι, πλησιάζουμε στο τέλος της θητείας μας και θα εργαζόμεθα μέχρι τα μέσα Απριλίου. Μετά από αυτά έχουμε τις ευρωεκλογέ προς το τέλος Μαΐου. Θα πρέπει να διεκπαιρεώσουμε όσο δυνατόν περισσότερα Δηλαδή ό,τι έχουμε μπροστά μας. Τις επόμενες λίγες εβδομάδες, αν θέλουμε να ψηφίσουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων τον Απρίλιο. Δεν είναι εύκολη η δουλειά που έχουμε μπροστά μας και ενώπιον σας, ενώπιον της Ρουμανικής Προεδρίας για πρώτη φορά στην ιστορία σας, συγχαρητήρια. Είμαστε πολύ ανοιχτοί για συνεργασία Καλωσορίζω τον Υπουργό, τον κύριο Άντων Άντων, Υπουργό Ενέργειας και τον κύριο Αλεξάνδρου Πετέσκου που είναι Υπουργό Επικοινωνίας και Κοινωνίας των Πληροφοριών. Ο Υπουργό Άντων υπεύθυνο για την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών θεμάτων. Για τα πάντα όσα αφορούν την ενέργεια, κάποιοι συνάδελφοι ίσως να τον ρωτήσουν και κάποιες ερωτήσεις για το κλίμα, διότι είναι στενά συνδεμένα η ενέργεια και το κλίμα. Και ο, ο Υπουργό ο κ. Πετρέσκου είναι υπεύθυνο για την πληροφορική και την ψηφιακή ατζέντα. Έχουμε το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη μπροστά μας. 9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η μελλοντική χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. τα διάφορα θέματα όσον αφορά την ενέργεια Αναμένεται πρόοδο από τον διαφόρων ζητημάτων επί Ρουμανική Προεδρία στο μέσο ηγεσία τη Ευρώπη, το Connecting Europe Facility, πολύ καλό. Κοινή κανόνε εσωτερική αγορά όσον αφορά το φυσικό αέριο. Πυρηνικό αφοπλισμό και ευρωπαϊκό εργαλείο για πυρηνική ασφάλεια. Ε, και διαφόρων των ελαστικών για την αποδοτικότητα και καύσιμα ο κανονισμό στην ενεργειακή απόδοση και ο κανονισμό για τη διακυβέρνηση ενεργειακή Ένωσης λόγω της απόσυρσης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση, στην περίπτωση της ψηφιακή ατζέντα και της, ε, των λογισμικών έχουμε επιτάπητο στο Connecting Europe Facility το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη η επανάχρηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Χθες ολοκληρώθηκε στις 6 το απόγευμα ή μάλλον στις 5 το απόγευμα, ολοκληρώθηκε το θέμα. Δεν έκρεμεί, αναμένει ψηφοφορία. Και Ευρωπαϊκή ε, Ασφάλεια και το κέντρο, τα διάφορα κέντρα για, το συντονισμό αυτών των θεμάτων. Έχουμε διάφορα θέματα, εννέα τον αριθμό. Ε, βέβαια, Εν τη αυτή περιπτώσει, στη συζήτηση με τους δύο υπουργούς της Ρουμανικής Κυβερνήσεως έχουμε νέα θέματα. Αγαπητοί φιλοξενούμενοι, αν επιτρέπετε να προτείνω κάτι. Ο Υπουργός ο κ. Άντων Άντων, αν έχει την καλοσύνη να ξεκινήσει τη συζήτηση, με την αρχική του παρέμβαση, μετά προτείνω να διεξαχθεί η συζήτηση και να δώσετε μετά απαντήσεις και μετά θα προχωρήσουμε και θα πάμε στο θέμα του ψηφιακού θεματολογίου και της ψηφιακής τεχνολογίας. Καλύτερα να διαχωρίσουμε τις δύο συζητήσεις. Ας ξεκινήσει λοιπόν τις συζητήσεις ο κύριος ε, Υπουργός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Μπούζεκ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παρουσία μου σήμερα εδώ, ενώπιόν σα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή ΣΥΤΡΕ, με σκοπό να παρουσιάσω τις προτεραιότητε της Ρουμανικής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμεινο του 2019, αποτελεί μια ιδιαίτερα μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδίως εσά, ε, Πρόεδρε Μπούζεκ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να παρουσιάσω το πρόγραμμα της ε, Ρουμανίας για το επόμενο εξάμεινο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης ε, τις προηγούμενες Προεδρίες. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τα επιτεύγματα της Αυστριακής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί τη φωνή των πολιτών και έναν από τους πιο μεγάλους πρόθητες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου. Επίσης, αποτελεί ουσιαστικό εταίρο για την Προεδρία στη διαδικασία ολοκληρώσης νομοθετικών φακέλων, πράξεων που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών για τα επόμενα έτη. Θα θέλαμε λοιπόν να αναπτύξουμε μια επικοδομητική συνεργασία τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ρουμανία συνειδητοποιεί την ευθύνη της εντολής που αναλαμβάνει καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή της εξέλιξής της. Επομένως, η Ρουμανική Προεδρία θα αναλάβει ένα ρόλο διαμεσολαβητή στην περίοδο της Προεδρίας προκειμένου να συνεισφέρει στην ε, ενοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης ε, και των κλιματικών πτυχών. Η Ρουμανία κατανοεί το διαμεσολαβικό, το διαμεσολαβικό αμερόληπτο ρόλο της ε, καθώς εκτελεί την εντολή της σε μια δύσκολη συγκυρία η σημερινή κατάσταση των φακέλων θέτονται σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο φιλοδοξία στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και την όθηση της Ευρωπαϊκή, του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου σε αυτή την εντολή. Στο πλαίσιο αυτών των προκλήσεων, η Ρουμανία, σε διάλογο με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, επιβεβαίωσε το γεγονό ότι η Ρουμανική Προεδρία θέλει να συνεισφέρει σημαντικά στην πολιτική σύγκληση και συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους τους πολίτες των κρατών μελών. Η αύξηση του πέδου συνοχής των κρατών μελών προκειμένου να υλοποιηθεί μια πιο ασφαλής Ευρώπη αποτελεί ένα στοιχείο για την εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την παγίωση του παγκόσμιου ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου στη συνέχεια να σας κάνω μια γενική παρουσίαση του προγράμματος της Ρουμανικής Προεδρίας βάση τριών πυλώνων η Ρουμανική Προεδρία ε, θέλει να επιδιώξει την κοινωνική και οικονομική συνοχή μέσω της προώθησης των θετικών αποτελεσμάτων ανθεκτικών πολιτικών ενέργειας ε, μέσω της επίτευξης στόχων προτεραιότητας σε σχέση με τις πηγές ενέργειας και την κλιματική αλλαγή και προωθώντας τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να προστατεύσει και να αναπτύξει την κοινή ενεργειακή αγορά, καθώς και τη χρηματοδότηση ζωτικών σχεδίων υποδομής. Όλες αυτές οι προσπάθειες είναι απαραίτητε για να πετύχουμε το στόχο του να έχουμε τον εφοδιασμό με μια ανταγωνιστική και βιώσιμη ενέργεια για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό δεν αρκούν μόνο οι ενεργειακές πολιτικές, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να δούμε και την υποδομή σε ό,τι αφορά το ψηφιακό επίπεδο, τις τεχνολογίες μεταφορών και τα κονδύλια για την έρευνα, αλλιώς και την ασφάλεια στον ενεργειακό αφαιδιασμό. ο πολίτης και το κάθε κράτος μέλος βρίσκεται στο επίκεντρο των κοινών μας προσπαθειών και ε, θέλουμε να επικεντρώσουμε στο προσπαθήθειά μας ε, στον ενεργειακό, στην ασφάλεια του ενεργειακού αφοδιασμού και στο να έχουμε προσιτές τιμές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα είναι εταίροι μας ε, στην επίτευξη του στόχου αυτού. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενέργεια. Έχουμε ομοδοποιήσει τις προτεραιότητές μας σε δύο θεματικές. Ε, καταρχήν, να συνεχίσουμε την περαιτέρω εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης, ε, της νομοθετικής διάστασης δηλαδή, και δεύτερον, ε, το μέλλον του ενεργειακού στήματος στην, στην Ενεργειακή Ένωση, δηλαδή με νομοθετική πτυχή. Αναγνωρίζουμε τη σημασία συνεχούς προσπάθειας για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση στην εφαρμογή των πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρουμανική Προεδρία θα ασχοληθεί με την νομοθετική διάσταση. Από την αρχή της θητείας μας δώσαμε πολύ μεγάλη προσοχή στην επιβεβαίωση πολιτικών συμφωνιών για το είδεσμι μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Εκτιμούμε τις δραστηριότητε της Αυστριακής Προεδρία προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως γνωρίζετε, η πολιτική συμφωνία που πετύχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του τελευταίου τριλόγου στις 18 Δεκεμβρίου επιβεβαιώθηκε την περασμένη εβδομάδα συνεδρίαση της Κορεπέρ στις 18 Ιανουαρίου και για την οδηγία αλλά και για τον κανονισμό σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά ενέργειας. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε τη θέση σε ισχύ αυτών των δύο νομοθετημάτων το συντομότερο. Σε ό,τι αφορά τώρα την οδηγία για το φυσικό αέριο, η Ρουμανική Προεδρία ε, δράει επικοδομητικά για τη διαπραγμάτευση του φακέλου αυτού. Επιθυμούμε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο διαφανές, έχοντας ε, κατά νου την πολιτική βούληση των συνομοθετών. Η Ρουμανική Προεδρία ξεκίνησε τις συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο την περασμένη εβδομάδα, στις 15 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας Ενέργεια. Αυτό το θέμα είναι πολύ λεπτό από πολιτική σκοπιά και υπάρχουν διαφορές απόψεις στα κράτη-μέλη. Η Ρουμανική Προεδρία κατανοεί ότι ο φάκελος αυτός αποτελεί προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα είναι φιδωλή προσπαθειών στο Συμβούλιο για την πρόθεσή του η Ρουμανική Προεδρία θα προωθήσει τις πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις στον κανονισμό σε ό,τι αφορά την ειδικοποίηση των ελαστικών ε, και το κανονισμό που αφορά την ενεργειακή διακυβέρνηση για τον Brexit. Στο πλαίσιο του Brexit αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι ο κανονισμό για την ετικετοσία των ελαστικών για τον ιδιωτικό τομέα και του καταναλωτέ. Η πρόθεσή μα είναι να σημειώσουμε ταχεία πρόοδο για να έχουμε μια γενική προσέγγιση σε αυτό το θέμα και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει μαζί σα το συντομότερο, αν το επιτρέψει, ο χρόνος σε ό,τι αφορά την προσαρμογή της οδηγίας ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα και του κανονισμού, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή διακυβέρνηση στο πλαίσιο του Brexit. Αναγνωρίζουμε την τεχνική φύση του φακέλου αυτού. Θα πρέπει με προτεραιότητα να το συζητήσουμε στην προοπτική του Brexit. Κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας, οι δύο ήδη είχαν άτυπες επαφές. Δεσμευόμαστε να φτάσουμε σύντομα σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά αυτό το σχέδιο. Το Συμβούλιο θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιβεβαιώσει τη διαπραγματευτική εντολή. Συντοποιούμε την ανάγκη να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον ενεργειακό τομέα, τομέα με υψηλή αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στι διοργανικέ διαπραγματεύσει σε σχέση με τον κανονισμό που αφορά το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη. Ο φάκελος αυτός ε, ε, είναι αντικείμενο διαχείρισης μαζί με τους τομείς μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Εκτιμούμε τις προσπάθειες της Αυστριακής Προεδρίας και τη γενική προσέγγιση που πέτυχε στο φάκελο αυτό στο Συμβούλιο Μεταφορών της 3 η Δεκεμβρίου 2018. Ο δικό μα στόχο είναι να, έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στι διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπω γνωρίζετε, ο πρώτο τριμερή διάλογο έλαβε χώρα χτε στι 22 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε με θετική έκβαση, ε, καθώ έχουμε περιορισμένο χρόνο προτείνουμε να έχουμε επικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας κατά νου ότι ο σκοπός αυτού να συμπίπτει με το στόχο της Ρουμανικής Προεδρίας, δηλαδή να έχουμε μια εύκολη μετάβαση από τη σημερινή περίοδο χρηματοδότησης του μηχανισμού στην μετέπειτα περίοδο από το 2021 και πέρα κατόπιν των πρώτων ανταλλαγών εντός του Συμβουλίου Ενεργείας το Δεκέμβριο θα οργανώσουμε ε, εις βάθος συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών ε, σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για ένα καθαρό πλανήτη. Πυλό φιλόδοξη στόχη για την ενέργεια και για τι ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα όπως τέθηκαν για τον ορίζοντα 2030 αποτελούν ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρίας για την μακροπρόθεσμη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Ξεκινώντας από το πλαίσιο αυτό, το όραμα της Επιτροπής αποτελεί μια χρήσιμη βάση για να συζητήσουμε τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ορίζοντα 2050. Έχουμε σχεδιάσει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο αυτό, στο, για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο ενέργεια και να υπάρχει μια συνεισφορά για τη Σύνοδο κορφή του Συμπίου στι 9 Μαου 2019. Η ενεργειακή κοινότητα είναι μία από τις ε, επιτυχίες της εξωτερικής ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει ε, εννιά συμβαλόμενα μέρη που συνεργάζονται προκειμένου να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην ενέργεια. Η Ρουμανία είναι ιδρυτικό μέλος της ενεργειακής κοινότητας από το 2005-2006 πριν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι αιτιολογείται το γεγονό ότι η Προεδρία της Ρουμανίας θα υποστηρίξει τις ε, δραστηριότητες της ενεργειακής κοινότητας. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε εντολή από το Συμβούλιο πέρσι το Νοέμβριο για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για να τροποποιήσει τη συνθήκη της ενεργειακής κοινότητας. Ο στόχος είναι να εντάξει μια σειρά προβλέψεων ως στοιχεία αμοιβαιότητας, υποχρεώσεις που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, Καθώ θα πρέπει να αποδεικτεί υποχρεωτική αξία μεταξύ των συμβολωμένων μερών τη ενεργειακή κοινότητα και των κρατών μελών τη Ένωση. Οι διαπραγματεύσει ξεκινούν τον Ιανουάριο Φέτο! και ελπίζουμε να ολοκληρωθούν το συντομότερο για να πετύχουμε τη Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς και την ασφάλεια του ενεργειακού εφηδιασμού. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μη νομοθετική διάσταση, η Προεδρία θα προτείνει μία συζήτηση για το μέλλον του ενεργειακού συστήματος στην Ενεργειακή Ένωση, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ενεργειακή μετάβαση και να πετύχουμε τους στόχους ε, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θέλουμε να θετήσουμε ένα σύνολο συμπερισμάτων Συμβουλίου για το θέμα αυτό τον Ιούνιο στο Συμβούλιο Ενέργειας. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών, λύσεων αποθήκευσης και νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Τώρα, επανερχόμενο στην νομοθετική διάσταση σε ό,τι αφορά τους φακέλους που αφορούν τον προπλισμό των πυρηνικών εργοστασίων, συνεχίζουμε τις προσπάθειες της Αυστριακής Προεδρίας για να βρούμε κάποιες συνενετικές λύσεις σε επίπεδο ομάδας εργασίας σε ό,τι αφορά τα τομικά ζητήματα. Το πρόγραμμα του παροπλισμού αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας για μία πιο ασφαλή Ευρώπη, παγιώνοντας την πυρηνική ασφάλεια και συνεισφέροντας στην προστασία του πολίτη και του περιβάλλοντος. Στο σημερινό πλαίσιο, όπου έχουμε προκλήσεις που τα κράτη-μέλη και οι άλλοι ε, διεθνείς παράγοντε αντιμετωπίζουν, η Προεδρία θα υιοθετήσει συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με την παγίωση τη ε, ε, πυρηνική ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά τι ε, συνεδριάσεις του Συμβουλίου θα λάβουν χώρα στις 4 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και στις 25 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Η Υπουργική Συνεδρία στις 4 Μαρτίου θα ασχοληθεί με νομοθετικά θέματα και στον, τον Ιούνιο θα έχουμε την οθέτηση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το ενεργειακό σύστημα της Ένωσης. Οι συνεδριάσεις θα δώσουν τον απαραίτητο χρόνο για τη συζήτηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την καθαρή ενέργεια και, τις συστάσεις, και των συστάσεων της Επιτροπής σε σχέση με τα εθνικά ολοκληρωμένα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Όπως βλέπετε αγαπητοί φίλοι, ο καιρός περνάει σε 45 λεπτά. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με δύο άλλους υπουργού από τη Ρουμανία. Λοιπόν, αν θέλετε να τελειώσουμε στις 3.45 πρέπει να συζητήσουμε και τα δύο ζητήματα μαζί. Και την ενέργεια και την πληροφορική. Και την ψηφιακή Ευρώπη. Μαζί. Αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, να ζητήσω τον κύριο Πετρέσκο να μας παρουσιάσει τώρα την δική του την άποψη για την Ρουμανική Προεδρία και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βόζεκ. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας πολλούς ευρωβουλευτές που πολύ ευγενικά μας έδωσαν χρόνο από το πρόγραμμα τους ε, για να τους συναντήσουμε χτες, προχτές και σήμερα. Και σας ευχαριστώ όλους για τα μεγάλα επιτεύγματα αυτά για το ότι εγκρίνατε πολλές από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ψηφιακής ενίας αγοράς και χάρη σε εσά έχουμε εγκρίνει τα δύο τρίτα του νομοθετικού πακέτου κομμάτι της ε, ψηφιακής εσωτερικής αγοράς ε, και βεβαίως η εντολή του Πρόεδρου είναι να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα νομοθετήματα και θα ήθελα να σπαταλήσω μόνο 7-8 λεπτά από τον χρόνο σας για να σας παρουσιάσω τις ε, αρχές ε, και τους στόχους ε, της Ρωμανικής Προεδρίας στον ψηφιακό τομέα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για όλη τη δουλειά που κάνετε σε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και να παρουσιάσω τις ε, προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Επιπλέον θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω τις προτεραιότητες μας στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και της ε, καινοτομίας του πολιτισμού και ακριβώς θέλουμε να υπάρξει μια συνεισφορά και προσθέμενη αξία στις προτεραιότητες και φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιοποίηση όλων των πτυχών της ζωής μας και της οικονομίας. Ε, το σύνθημά μας είναι μια Ευρώπη, μια ψηφιακή Ευρώπη χωρίς ε, σύνορα. Γιατί μόνο έτσι η Ευρώπη θα είναι ισχυρή και ανταγωνιστική. Χρειαζόμαστε ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες θα είναι διαλειτουργικές, ε, φιλικές προς τον χρήστη, θα μειώνουν τα κοινωνικά χάσματα και θα έχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες θα είναι σχεδιασμένες σήμερα με τις ανάγκες των πολιτών, της βιομηχανίας, της κοινωνίας και της οικονομίας σε συνεργασία και με γειτονικέ χώρες ε, για μια πιο ισχυρή ασφαλή ανταγωνιστική Ευρώπη. Προσβασιμότητα για όλους, ειδικά για τις περιοχές της υπαίθρου, υπηρεσίες, υποδομές ε, και νέες δουλειές. Οι προτεραιότητε ε, της Προεδρίας μας ε, πάνε σε τέσσερι κύριε γραμμές. Καινοτομία, κυβερνοασφάλεια, ηλεκτρονικέ δεξιότητε και γυναίκε στην τεχνολογία. Όλα αυτά εξαρτώνται από την ικανότητα τη Ευρώπη να εντείνει τη χρήση προχωρημένων τεχνολογιών, όπω το blockchain, η πέμπτη γενιά και της τηλεφωνίας, ε, και αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και των ψηφιακών ικανοτήτων της η Ρουμανική Προεδρία θα εστιάσει την δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για τις ε, καινούριες εταιρείες, ε, έτσι ώστε κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη να ωφελείται από την ψηφιακή καινοτομία για να υιοθετηθούν ε, και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα δεδομένα από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Θα κοιτάμε προς το μέλλον και τέτοια θα είναι και η προσέγγιση μας για τις νέες ε, τεχνολογίες. Δίνουμε ε, υψηλή προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια, καθώς έχει σημασία για την προστασία των στρατηγικών συμφερόντων μας και να μπορέσουν οι πολίτες μας να ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Πρέπει να έχουμε μηχανισμούς ε, κυβερνοασφάλειας, και κυβερνοάμυνα για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την εξέλιξη της ψηφιακή ε, οικονομίας ε, διασφαλίζοντας ε, τις εταιρείε και τις υποδομέ που διατηρούν την οικονομία και την δημοκρατία μας. Θα πρέπει να αποφύγουμε την διαρροή εγκεφάλων για να μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή ψηφιακή εικόνα. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε ψηφιακές δεξιότητες για να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, για να αυξηθεί η ποιότητα ζωής, να μπορούν όλοι οι πολίτες να ωφεληθούν από, την από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα καθώς οι προκλήσεις αυτές κινούνται πάρα πολύ γρήγορα και απαιτούνται νέες ή προχωρημένες δεξιότητες για την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν μεγάλη σημασία αυτές, ιδιαίτερα για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για το ψηφιακό οικοσύστημα το οποίο θα ευνοήσει την καινοτομία και τις νοοφυεί επιχειρήσεις. Γι' αυτό η Προεδρία μας ε, θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην αύξηση της, ε, του ψηφιακού αλφαβητισμού στην Ευρώπη, την αύξηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, προώθηση των ε, ταλέντων, της δημιουργικότητας στην κυβερνοασφάλεια και στις σχετικές τεχνολογίες. Το δυναμικό ρουμανικό ψηφιακό πνεύμα φαίνεται στην πράξη και στο πρόγραμμά μας για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα εργαστούμε προς την πρόθεση περισσότερων γυναικών στον τομέα της ε, τεχνολογίας έτσι ώστε τα κορίτσια και οι γυναίκες να έχουν υπόψη τους τις νέες ψηφιακές θέσεις εργασίας. Όλοι οι νομοθετικοί φάκελοι επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική, και θα έχουμε μεγάλη φιλοδοξία για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε όλους. Οι νομοθετικοί φάκελοι έχουν ένα κοινό στοιχείο δηλαδή τα δεδομένα τα οποία θα δημιουργούν σημαντική προσθέμενη αξία αλλά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα να μπορέσουμε ακριβώς να τα χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο για να ωφεληθεί η οικονομία και η κοινωνία. Όλα τα πολιτικά και νομοθετικά μέτρα να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε καινοτόμες τέτοιες τεχνολογίες και θα αυξήσουν την αξία της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας των δεδομένων σε 700 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020 και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσο δυνατόν περισσότερο ως σημαντικό κομμάτι της καινοτομίας. Ο δημόσιος τομέας είναι ένας τομέας έντασης δεδομένων, οπότε η χρήση αυτών των δεδομένων μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών, στην ανάπτυξη της ε, τεχνητής νοημοσύνης ε, στην έρευνα των ανοιχτών δεδομένων και να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά προβλήματα π.χ. στην υγεία ή τις ε, μαζικές μεταφορές. Επιτύχαμε χτες μια προσωρινή πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναθεωρημένη οδηγία για τα δεδομένα του δημοσίου τομέα. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ευρώπη για να αυξηθεί η διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες και για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης επίσης συνεισφέρει περαιτέρω στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτές τις ε, τεχνολογίες. Για να επιτύχουμε όλα αυτά τα ανωτέρω σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε φιλόδοξες επενδύσει, ειδικά όταν μιλάμε για του υπερυπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, κύβερνο ασφάλεια και προχωρημένε ψηφιακέ δεξιότητε και να υπάρχει μια ευρεία χρήση από τι επιχειρήσει και τον δημόσιο τομέα, αλλά και σε σχέση με την ανάπτυξη μια σωστή ψηφιακή υποδομή. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε το δυνατόν περισσότερο στο πρόγραμμα ψηφιακή Ευρώπη και στο μέσο συνδέοντα την Ευρώπη. Μια άλλη σημαντική προτεραιότητα της ε, Προεδρίας μας. Για να μπορούμε λοιπόν να ανταγωνιστούμε παγκοσμίω, η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύει στις πιο προχωρημένες ε, τεχνολογίες, στην έρευνα και στην καινοτομία, διασφαλίζοντας την διαλειτουργικότητα και την βέλτιστη χρήση. Μια πραγματικά εσωτερική ψηφιακή και ενιαία αγορά σημαίνει ακριβώς δημιουργία αξίας, ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας ε, και της εμπιστοσύνης την δημιουργία ψηφιακών κόμβων καινοτομία επιπλέον. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην νομοθετική πρόταση για τα κέντρα αριστείας κυβερνοασφάλειας και έρευνας. Θέλουμε να προχωρήσουμε στο δυνατόν περισσότερο στις διαπραγματεύσεις του συγκεκριμένου θέματος. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της ε, κυβερνοασφάλειας τις ε, τεχνολογικές ικανότητες που είναι απαραίτητες και θα ενισχύσει την πολιτική προσέγγιση μας στο θέμα για καλύτερη συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα τοπίο το οποίο εξελίσσεται ραγδαία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το θέμα αυτό για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Από την τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας του 2009 οι ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και όλο και περισσότερο πλέον οι κοινωνίες ε, και οι οικονομίες μας βασίζονται σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω διαδικτύου όπως ε, τα μηνύματα και ε, οι φωνητικές κλήσεις μέσω IP κτλ. Λοιπόν η Προεδρία μας ξεκινάει ήδη από τη συμφωνία στο Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2018 και σκοπεύουμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που μας συνάντησαν πριν από τη συνεδρίαση αυτή και σε όσους συνεισέφεραν στα εξαιρετικά επιτεύγματα μέχρι στιγμής και να σας πω ότι είμαι πάντα στην διάθεσή σας όποτε θέλετε να συζητήσουμε όλοι μαζί ή τέτα για να είναι η Προεδρία μας επιτυχής. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Τώρα πάμε στη συζήτηση. Οι συντονιστές μας, οι εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων πρώτα απ' όλα. Ένας από κάθε πολιτική ομάδα, εκ μέρους του ΕΛΚ, ο συνάδελφος Έρερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργοί, που ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Υπό το φως της ελλείψεως χρόνου θα ήθελα να μειώσω τις ερωτήσεις μου σε δύο. Καταρχάς, σωστά αναφερθήκατε στη σημασία της κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο το αμυντικό. Πώς αντιλαμβάνεστε την πρόταση του Κοινοβουλίου, έχουμε την ΕΝΙΣΑ, που δεν είναι εκτελεστικός φορέας με την κλασική έννοια του όρου. Αφορά διάδραση, ανταλλαγή πληροφοριών κλπ. Ανανέωσε την πρότασή του όμως το Κοινοβούλιο. Από το πρόγραμμα έρευνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να πάρουμε ένα ποσό για να το δώσουμε στις οργανώσεις για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, όπως είναι η Europol. Έχουμε 250 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα για την κυβερνοασφάλεια, για το ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά ο προπολογισμό για τη Europol είναι 5 εκατομμύρια ευρώ για επιχειρησιακό κομμάτι ή επιστημονικό και τεχνολογικό κομμάτι. Θα ήταν συνετό να μεταφέρουμε πόρους από το πρόγραμμα έρευνας και ασφάλειας που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ πιο επιφανείς οργανισμού θα λέγαμε, πιο συγκεκριμένου. 5 εκατομμύρια ευρώ που εν συγκρίση με τα 250 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι τίποτα αυτά που διαθέτουμε για την έρευνα. Αλλά είχε μπλοκαριστεί το ποσό από το Συμβούλιο. Άλλη ερώτηση που αυτή σχετίζεται με το ψηφιακό πρόγραμμα αλλά και το πρόγραμμα το ερευνητικό. Πάντα μιλούμε για συνέχεια. Οι συμπράξεις, οι τερκές σχέσεις, αυτές οι συμπράξεις που συνδέονται ε, με την πληροφορική, όπως το Photonics, που ήταν η πιο καλά βαθμολογημένη σύμπραξη. Είχε πει ότι σε επιτροπολογία θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις μετά το 2020 και το Συμβούλιο αοριστολογεί. Αναφέρει συνέχεια, αναφέρεται στους τομείς της σύμπραξης. Δεν γίνεται όμως λόγος για εφιστάμενες συμπράξεις, όπως το Photonics. Είναι, ε, ε, καλύπτει την αεροναυπηγική λοιπά ο τομέας των φωτονίων. Αλλά δεν εμφανίζεται πουθενά στη θέση του Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε κάποια ελευθερία για να αποκαταστήσουμε τους διάφορους φορείς και πώς θα χρηματοδοτηθούν, αλλά χρειαζόμαστε και διαβεβαιώσεις από τη βιομηχανία, ότι συνεχώς χορηγούνται τα χρήματα σε αυτούς τους τομείς. Ερώτηση. Βλέπετε το σχεσισμό μεταξύ του ψηφιακού πακέτου και του ερευνητικού προγράμματος. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, εκ μέρους των ο κύριος Νίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο υπουργού, τον κύριο Αντών και τον κύριο Πετρέσκου. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε την οδό που ξεκινήσατε γιατί μόνο 3,5 μήνες έχει δυστυχώς τη διαθεσή η Προεδρία, όχι 6 μήνες όπως έχουν άλλες Προεδρίες. Είναι πολύ μεγάλες οι προσδοκίες γιατί είναι πολύ σημαντική η φάκελη αυτή και ταυτόχρονα είμαστε και σε προκλογική περίοδο και αυτό δεν θα σας βοηθήσει και πολύ. Όμως ε, βασίζομαι πάρα πολύ ε, στο πολύ καλό οργανωτικό πνεύμα και μαχητικό πνεύμα που έχετε. Θέλω να αναφέρω δύο πράγματα. Καταρχήν βρίσκεστε στην Επιτροπή Ήτρε Πρόκειται για τη, μία από τις ε, πιο σημαντικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολείται σχεδόν ε, με όλα όσα έχουν να κάνουν με την οικονομία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη. Είναι μια τεχνική επιτροπή η οποία έχει κατορθώσει, υιοθετήσει πάρα πολλούς φακέλους, πολύ σημαντικούς για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, λεχθέντος αυτού. Έχω ε, μια πρώτη παράκληση για τον κύριο Αντών ε, να εξετάσετε πολύ προσεκτικά την οδηγία για το φυσικό αέριο. Είναι μια οδηγία που την εθετήσαμε στην Ήτρε και αγωνιστήκαμε <coughs> πολύ γιατί από την υιοθέτηση αυτής της οδηγίας εξαρτάται η διασφάλιση μιας ευρωπαϊκής αγοράς που να είναι αποτελεσματική για να έχουμε και ένα καλύτερο ανταγωνισμό και πιο καλές τιμές που θα πληρώνουν οι πολίτες μία αγορά όπου θα έχουμε διαφοροποίηση των πηγών αφοδιασμού και αυτό θα επιτρέψει ασφάλεια στον εφοδιασμό. Ξέρετε, καθώς είστε από τη Ρουμανία, όταν κάνει πολύ κρύο, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν δεν έχεις από πού να πάρεις αέριο και υποφέρει όλη η περιοχή και πόσο νόημα έχει να έχουμε διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού. Δυστυχώς έχει τελματώσει αυτή η οδηγία. Στο πρώτο εξάμεινο το προηγουμένό τους ε, είχε τελματώσει. Και θα ήθελα να μου πείτε τι προσπάθειες θα κάνετε για να υιοθετηθεί η οδηγία αυτή υπό τη δική σας προεδρία. Τώρα, για τον κύριο Πετρέσκου, την ερώτηση για την κυβερνοασφάλεια. Και εμείς αγωνιστήκαμε πολύ εδώ για να ενταχθούν και τα κριτήρια και τα στοιχεία που να βελτιώσουν την καταπολέμηση της πειρατείας. Όμως αυτό το κέντρο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πιστεύετε ότι θα πρέπει ε, να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή ποιο θα είναι αυτό το χαρακτηριστικό που να μας δίνει τη διασφάλιση ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχουμε ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και αυτό το περιμένει πάρα πολλοί κόσμο. Θέλουμε να έχουμε ένα ασφαλή κόσμο. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τι επιγραμμικέ υπηρεσίε ή τα κινητά μα. Απλώ θέλουμε να ξέρουμε ότι είναι ασφαλή αυτά και δεν εκτίθεται ε, σε επιθέσει από διάφορου hacker που θα πρέπει να τι ε, καταπολεμούμε και μέσω μια κοινή προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Ο κ. Τέσακ. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. E, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήσατε επίσης για την χρήση των δεδομένων του δημοσίου τομέα. Κύριε Πετρέσκου, είπατε πως ε, κατά τη διάρκεια της ε, Ρουμανικής ε, Προεδρίας σκοπεύετε να εργαστείτε περαιτέρω στην πέμπτη γενιά κινητής τηλεφωνίας και μιλήσατε για την προετοιμασία μιας διάσκεψης το 2019 και η Κομισιόν εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό και Ακριβώς ε, το ζήτημα είναι να εμφανιστεί ενιαία η Ευρωπαϊκή Ένωση και ενωμένη στην διάσκεψη του ΟΗΕ. Έχω λοιπόν μία ερώτηση. Θεωρείτε ότι προγραμματίζονται κάποιοι περιορισμοί στους προμηθευτές ε, τελικών ε, συσκευών και πώς προετοιμάζεται η Προεδρία για την επεξεργασία μιας κοινή στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπατε κάτι πράγματα, αλλά θα ήθελα λίγο να επεκταθείτε. Τώρα, για την προετοιμασία της ε, διάσκεψης ε, για την ε, τεχνητή νοημοσύνη στην οποία εργάζομαι. Υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Μία άλλη ερώτηση. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την ανατολική γειτονία. Θα υπάρξει οπωσδήποτε ένα επίσημο συμβούλιο μαζί με την Ανατολική Γειτονία το Μάρτιο στην, στο Βουκουρέστι και θα έχουμε εκεί πέρα εκπροσώπους των κρατών μελών και των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας και θα υπογραφεί μια συμφωνία για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Σε ποια κατεύθυνση θα πάει αυτή η εναρμόνιση και σε ποιους ε, κλάδους τι στόχους ε, έχετε. Η ανατολική γειτονία είναι πάρα πολύ σημαντική και ακριβώς θέλουμε η ανατολική αυτή αγορά να γίνει προσβάσιμη. Και τώρα για το φάσμα και τα τέλη περιαγωγής ε, έχει μεγάλη σημασία αυτό, δηλαδή η ασφάλεια προγραμματισμού. Τέλος, τι σχέδια έχει η Προεδρία για την ψηφιακή Ευρώπη και οι προλαλήσαντες μίλησαν επίσης για τις ευρωεκλογές τον Μάιο μπορείτε να μας πείτε αν θα υπάρξει κάποια ψηφοφορία στο Κοινοβουλίο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μιλνερέ, από την άλλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς που ήρθαν. Θα είμαι και εγώ σύντομη. Θα εστιαστώ επί θέματος που είναι βασικό μου θέμα Είμαι συγγήτρια για το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη. Μαζί με του συναδέλφου εργαζόμαστε σκληρά. Και καταλήξαμε τελικά σε καλό αποτέλεσμα. Όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, Πετρέσκου, και επειδή τονίσατε τον ψηφιακό τομέα και την κυβερνοασφάλεια, και η κυβερνοασφάλεια ανήκει στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Ένα από, ένας από τους μεγάλους στόχους, από του πέντε στόχου που έχουμε. Οι, με ε, διάδοση της τεχνολογίας, τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Έχει επιβεβαιωθεί εντολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις από σήμερα. Βασικό εργαλείο για το πρόγραμμα, για την επιτυχία μάλλον του προγράμματος, θα είναι η δημιουργία του δικτύου ψηφιακής καινοτομίας, κόμβοι που θα διαδοθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Είναι κάτι χρονοβόρο για τα κράτη-μέλη. Και ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Θέλω να είμαι σίγουρη, βλέπετε, ότι πριν το τέλος της θητείας μας θα καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα και θα δώσουμε χρόνο στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν, να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό. Κάτι που αναμένεται από καιρού και είναι μια ευκαιρία. Αν έχετε την καλοσύνη, δώστε μου κάποια εικόνα. Τι εικόνα έχετε για αυτό το θέμα. Μπορείτε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες, σας παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου, δεν ακούμε. Uh, uh, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να υποβάλουμε ερωτήσεις. Η ερώτησή μου αφορά και το τέλος της θητείας της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου. Εδώ και ένα χρόνο περιμένουμε κάποιες εξελίξεις θετικές όσον αφορά ε, την οδηγία Είσαστε από τους πατέρες των συμβιβαστικών λύσεων που βρήκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, κυρίως αυτή η Επιτροπή. για την οδηγία, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να πείσει την πρώην ε, προεδρία, τις προηγούμενες προεδρίες να ασχοληθούν με το θέμα του φυσικού αερίου, της οδηγίας σχετικής. Χρειαζόμαστε τη νέα οδηγία, πιστεύουμε, και είμαι πεπισμένη ότι εργαστήκαμε επί μακρών επί που υπόσχονται πολλά. Έπρεπε να αναπτύξουμε το δικό μας ενεργειακό σχέδιο, ενεργειακά σχέδια και να βελτιώσουμε και την ασφάλεια την ενεργειακή. Έπρεπε να ανταποκριθούμε και στους στόχους μας για το κλίμα. Σε αυτό το πλαίσιο καλωσορίζω τη δική σας πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ Πετρέσκου διότι ανακοινώσατε ότι θέλετε να πετύχετε συμφωνία στο Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για το φυσικό αέριο. Η ερώτησή μου, θα μπορεί να γίνει αυτό πριν από τις ευρωεκλογέ και πριν το τέλος της θητείας. Θα μπορέσουμε να αποδείξουμε στους πολίτες μας ότι είμαστε ικανοί να βρούμε συμβιβασμό στο Συμβούλιο και ένα καλό τέλος για αυτή την υπόθεση διότι νομίζω ότι οι πολίτες όσον αφορά το θέμα έβρισκαν ξανά την απόδειξη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε σε θέση να βρούμε συμβιβασμούς επί των μεγάλων θεμάτων. Πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε ικανοί να δράσουμε και ότι υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δύσκολο τομέα ε, του φυσικού αερίου από την Ρωσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου. Ο κύριος Σιλικιώτης, εκ μέρους της ε, ΓΚΟΕ. Ήθελα να καλωσορίσω και εγώ και να ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ τους δύο υπουργού και την ε, ε, ενδιαφέρουσα παρουσία τους και τις θέσεις που έχουν θέσει. Ε, θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία και να εκφράσω τις ιδιαίτερες με ευχαριστίες στη Ρουμανική Προεδρία για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να καταλήξουμε χθε τη συμφωνία στον Τρίλογο για την αναθεώρηση τη οδηγία PSI για τα ανοιχτά δεδομένα και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του δημόσιου τομέα. Έχουμε πετύχει μια πολύ καλή συμφωνία, η οποία ε, μέσω τη νέα νομοθεσία δεν διασφαλίζει πω τα δεδομένα θα παρέχονται δωρεάν προ όφελο τη κοινωνία και θα αξιοποιούνται σημαντικά αυτά τα δεδομένα, τα οποία ε, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέες αναδυόμενες επιχειρήσεις θα βοηθηθούν πολύ από την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ε, και πρέπει να πω ότι ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο κ. Πετρέσκου έθεσε τα θέματα της ψηφιακής οικονομίας και εδώ στη συζήτηση είναι, είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει βήματα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή οικονομία και θεωρώ ότι η Ρουμανική Προεδρία μπορεί να βάλει το στίγμα τη αυτό το εξάμεινο για την ψηφιακή οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα ενέργεια, το πρόγραμμα τη Ρουμάνικη Προεδρία είναι βασική προτεραιότητα ορίζεται η ανάγκη ενίσχυση του ενεργειακού συστήματο, αξιοποιώντα τι νέε τεχνολογίε και βελτιώνοντα τι υποδομέ και τα συστήματα αποθήκευση. Αναφίβολα αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Άντων, Ωστόσο, η ανάγκη να επισημάνουμε πω σε πολλέ φορέ υπάρχουν υποδομέ, υπάρχουν τα δικτύα, υπάρχουν οι αγωγοί, αλλά τα νοικοκυριά αδυνατού δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να εγκαταστήσουν τα συστήματα που απαιτούνται για αξιοποίηση της φθηνής ενέργειας. Έτσι η παροχή ενέργειας στους δεν μπορεί να διασφαλιστεί ως ένα δημόσιο κοινωνικό και ανθρώπινο αγαθό. Ε, όταν λοιπόν μιλάμε για τη δημιουργία τη Ενεργειακή Ένωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε πω βασική προπόθεση είναι να στρίξουμε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που σήμερα υποφέρουν από την ενεργειακή φτώχεια. Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα σημαντικό θέμα, το έχουμε θέσει πολλέ φορέ εδώ στην Επιτροπή. Αλλά αυτό που αναμένουμε είναι να υπάρξει ένα. Ε, και αναμένουμε να συμβάλλει η Ρωμανική Προεδρία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για καταπολέμηση τη ενεργειακή φτώχεια που ταλανίζει εκατομμύρια συμπολίτε μα στην Ένωση. Ε, ο στόχο τη ε, δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτη στα προσόφερε των λαών. Και πρέπει να υπάρξει ένα κοινό ορισμό, ένα, ένα, κάτι που απασχολούμαστε εδώ και πολύ καιρό, για το τι είναι ενεργειακή φτώχεια μαζί με ένα σύνολο κριτηρίων ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την προτεραιότητα για για την οδηγία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να επισημάνουμε πω το πιο σημαντικό είναι να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερβεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην ενεργειακή τη ασφάλεια και στην ενεργειακή τροφοδοσία. Και θα ήθελα ακριβώ εδώ να επισημάνω ότι πρέπει να πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε την κυριαρχία των κρατών μελών, και αναφέρομαι ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, και τα ε, σημαντικά κοιτάσματα που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή είναι κοιτάσματα τη Ένωση και πρέπει να αξιοποιηθούν για την ενεργειακή ασφάλεια τη Ένωση. Ευχαριστώ. Thank Uh, so other speakers ομιλητές. Έχω ένα μακρύ κατάλογο από τους υπόλοιπους συναδέλφους που σου το λόγο. Θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Παρακαλώ, κύριος Τερσανόφσκι. Σε ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Σε ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Έχω μία ανακοίνωση και μία ερώτηση. Στον ε, κύριο Υπουργό, τον κύριο Άντων, ε, βρήκα ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπε για την ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας. Προς ποια κατεύθυνση θέλετε να γίνει η συζήτηση, γιατί συχνά βλέπουμε εδώ πέρα στην Επιτροπή πως είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Με ενδιαφέρει λοιπόν αυτό γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση σε ελαιόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ και τον κύριο Πετρέσκου. Σας συνάντησα και πριν και σας ευχαριστώ. Εγώ άκουσα την απάντηση που ήθελα πριν, αλλά... Θα ήθελα να σας, να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στους τρεις μήνες που έχετε για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε όλα τα ζητήματα νομοθετικά και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ernst. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, συγχαρητήρια που αναλάβατε την Προεδρία του Συμβουλίου και άκουσα πολλά θετικά πράγματα για την Ενεργειακή Ένωση και μια ερώτηση απευθύνω στον κύριο Άντων. Ε, γνωρίζετε πως υπάρχει μια περιοχή με άνθρακα και πολλές περιοχές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα απομακρυνθούμε σιγά σιγά από τον άνθρακα για οικολογικού λόγους. Χρειάζεται λοιπόν μια κοινωνική στήριξη. Οπότε το ερώτημά μου είναι ποιε ιδέες έχει η Προεδρία σα για την δίκαιη μετάβαση, την στήριξη των περιοχών ε, εκείνων που θα βρεθούν στην μετάβαση αυτή και θα πρέπει ή θέλουν να αλλάξουν μοντέλο, ποια θα μπορεί να είναι η βοήθεια και η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς ε, το βλέπετε, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην έρθει αυτή η αλλαγή επειδή δεν τη θέλει το Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ζωρίγιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργή. Βρίσκεται η Ρουμανική Προεδρία σε μια στιγμή μεγάλων προκλήσεων και δυσκολιών. Όμω υπάρχουν κάποιοι φάκελοι στους τομείς σας όπως η Ψηφιακή Ένωση και η Ενεργειακή Ένωση που μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα όπως ε, καθώς έχουμε περιορισμένο χρόνο θα περάσω κατευθείαν στις ερωτήσεις. Ποια βήματα θέλει να κάνει η Ρουμανική Προεδρία για να υλοποιηθούν αυτές οι δύο ενώσεις, η ενεργειακή και η ψηφιακή και συγκεκριμένα για να θέσετε ε, την, ε, τους όρους μετάβασης για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Γιγαμπάιτ. Επίσης, ε, για το πρόγραμμα ψηφικής Ευρώπης, ε, ε, η Ρουμανική Προεδρία ακόμη δεν έχει δέσει τον πρώτο τριμερή διάλογο. Εμείς δεν μπορούμε απλώ να σκεφτόμαστε θεωρητικά. Θα πρέπει να περάσουμε στην πράξη και ακόμη δεν έχουμε ορίσει την πρώτη τεχνική συνεδρίαση για το πρόγραμμα αυτό. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο εξή, ε, ότι υποστηρίζουμε τη Ρουμανική Προεδρία στην πρωτοβουλία Wi-Fi for You. Είναι ε, πάρα πολύ μεγάλη πρωτοβουλία και εγώ βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ, κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στη διευκόλυνση σύνδεσης ε, της Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο είχε διάφορες προτάσεις. Χθες ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Το Κοινοβούλιο έχει προτάσεις ε, σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση των ψηφιακών διαδρόμων. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψη της ε, Προεδρίας ε, για το θέμα αυτό. Γιατί υπάρχουν προτάσεις και από την Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο. Επίσης, το Κοινοβούλιο πρότεινε ένα πρόγραμμα πλαίσιο. Δηλαδή, πριν να ξεκινήσει ο μηχανισμός αυτός, η Κομισιόν παρουσιάσει ένα πρόγραμμα πλαίσιο που θα παρουσίαζε την προβλεψιμότητα και τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν πολύ πιο καλά σχέδια και προγράμματα. Θα ήθελα να ξέρω τη θέση της Ρουμανικής Προεδρίας για το θέμα αυτό. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφος Γιάβορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσω την ερώτηση της συνεδέλφου Ρεμπέκα Χάρμς για αυτή το θέμα της οδηγίας που συζητήθηκε επανειλημμένα μαζί σας από διαφορετική οπτική γωνία. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο θέμα ενεργειακό και ενεργειακής ένωσης ή κατών, όλα τα κάτι Μεσοευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζονται από τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Άρα και εταίροι μας στην ενεργειακή κοινότητα επηρεάζονται κατά πολύ από τα αποτελέσματα οδηγία για το φυσικό αέριο και τις σχετικές συζητήσεις. Ερώτηση προ τη Ρουμανική Προεδρία. Οι πτυχέ ενεργειακής ασφάλειας, οι διακοπές, στατηγική εταίροι κλπ. Πιστεύετε ότι οι πτυχέ αυτέ λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Λαμβάνονται υπόψη δεν είναι μόνο θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ευρύτερο. Καλύπτει και άλλε χώρε και μέλη τη ενεργειακή κοινότητα Η Ρουμανική Προεδρία μπορεί να επιταχύνει τις συζητήσεις στο Συμβούλιο για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των κρατών μελών και των χωρών που είναι μέλη της ενεργειακής κοινότητας. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος του καταλόγου ομιλητών. Υπάρχει άλλος. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Λοιπόν, αν επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, αναφερθήκανε στην αναθεώρηση οδηγίας στο φυσικό αέριο κάποιοι συνάδελφοι. Θεωρώ ότι είμαι υπεύθυνο γι' αυτό, σαν εισηγητή. Να πω ότι από την άλλη πλευρά είμαστε πολύ ανοιχτοί όσον αφορά ταχείε και επικοδομητικέ διαπραγματεύσεις και θέλουμε να πετύχουμε το βασικό στόχο της αναθεωρήσεως που είναι προφανέστατο. η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα και μετά θα πρέπει να καλυφθούν και ανησυχίε που εξέφρασαν τα κράτη-μέλη. Οι φυστάμενε υποδομέ Φερρυπίν, είναι συγκεκριμένο πρόβλημα, γνωστό. Το θέμα των ανάντι ε, αγωγών, ε, μετακύληση αρμοδιοτήτων και η εφαρμογή των διαφόρων κωδικών ε, των δικτύων. Ίσως και κάποιες άλλες πτυχές που θα μπορούσαν να συζητηθούν. Πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αν οι διαπραγματεύσουν, δεν επιτυγχάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε καμία συζήτηση. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ και τους δύο υπουργού να απαντήσουν στις τεθείς ερωτήσεις και να προβούν στα καταληκτικά τους σχόλια. Ορίστε. Α, κάτι στα γρήγορα, μια διόρθωση. Όταν μίλησε για την καθυστέρηση στο πρόγραμμα του τεχνικού τριμερούς διαλόγου στην, ε, για την ψηφιακή Ευρώπη δεν ήταν τεχνικός διάλογος, μιλούσα, εννοούσα τον πολιτικό διάλογο, όχι τον τεχνικό, τον πολιτικό. Αυτή είναι η διόρθωση. Σας ευχαριστώ. Όπως αναμενόταν, διαπίστωσα ότι οι περισσότερες ερωτήσεις αναφέρθηκαν ε, στην οδηγία για το φυσικό αέριο. υπό την ιδιότητά μας ε, από τη θέση της Προεδρίας. Όπως σας είπα, εμείς εφαρμόσαμε όσα ζητήθηκαν στο Συμβούλιο της 21ης Δεκεμβρίου, δηλαδή μια ταχεία προσέγγιση αυτής της προβληματικής. Συνεπώς, στις 15 Ιανουαρίου θέσαμε στη συζήτηση ένα νέο κείμενο σε όλα τα κρατημέλη και ήδη στην Τεχνική Επιτροπή και ήδη λάβαμε κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με το κείμενο αυτό. Τώρα είμαστε σε θέση βάσει των ετοιμάτων των κρατών μελών να προσαρμόσουμε το κείμενο τα οποίο θα παρουσιάσουμε και στη συνέχεια. Η δική μας επιθυμία είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος, για όλα τα κράτη που γειτονεύουν μαζί μας και ενδιαφέρονται για την οδηγία αυτή. Αυτή η οδηγία είναι η επιθυμία να φτάσει γρήγορα σε τριμερή διάλογο για κατόπιν να ληφθούν οι αποφάσεις. Έχω ξανακάνει τη δήλωση αυτή και την ξανακάνω, αλλά επαναλαμβάνω. Είναι η βούληση, η εκπεφρασμένη βούληση όλων των κρατών μελών Είναι ένα πολύ καυτό θέμα σήμερα, το οποίο συνεχώς το συζητάμε. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι έτοιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συζήτηση. Εμείς θέλουμε η Προεδρία να κάνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και στο χρόνο που μας απομένει να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την οδηγία αυτή. Επίσης, θα ήθελα να σας πω το εξή. δεν το είπα στην αρχή, αλλά μπορεί να Α, είδατε στην παρουσίασή μου ότι και στις 4 Μαρτίου έχουμε προγραμματίσει συμβούλιο και τον Ιούνιο. Το Συμβουλίο της 4ης Μαρτίου θα συζητήσει τα προβλήματα που θέλουμε να επιληθούν μαζί με το Κοινοβούλιο. Προτείναμε όμως αυτό το πρόσθετο συμβούλιο, γνωρίζοντας ε, ότι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας ε, είναι περιορισμένος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ότι έχουμε προβλήματα στον τομέα των πυρηνικών. Όμως ήθελα να σας πω ότι τόσο συζητήσαμε δεν σημαίνει ότι θα τροποποιήσουμε την οδηγία. Ίσως αυτό να έχει να κάνει με την έννοια των όρων. Μας ενδιαφέρει το θέμα της ασφάλειας των πολιτών. Μας ενδιαφέρει το θέμα της ασφάλειας των υλικών δεν θέλουμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη οδηγία, η οποία είναι πολύ αυστηρή και αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Και τέλος, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κ. Σιλικιώτης. για την ενεργειακή ανέχεια. Η ενεργειακή ανέχεια είναι πρόβλημα και είναι πρόβλημα όλων μας. Σε κάποιες χώρες ίσως να είναι πιο έντονο το φαινόμενο από κάποιες άλλες. Όμως, αποτελεί μέρος της στρατηγικής που θέλουμε να αναπτύξουμε. Και βρίσκεται στο στόχαστρο της Προεδρίας μας. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που υπογραμμίσατε τα πιο σημαντικά θέματα και για τις παρατηρήσεις σας. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πετρέσκου για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Χαίρομαι που υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τον ψηφιακό τομέα και πολλές ερωτήσεις απευθύνθηκαν σε μένα. Οπότε προφανώς έχουμε μια πολύ καλή διασυνδεδεμένη προσέγγιση. Ένα καλό σημάδι αυτό. Και θα εκμεταλλευτώ την καλοσύνη σα που μου δίνετε χρόνο. Ε, ζητώ συγγνώμη αν δεν ακολουθώ ακριβώς την σειρά των ερωτήσεων. Θα προσπαθήσω όμως ε, να απαντήσω με τρόπο συνθετικό τις περισσότερες ερωτήσεις και αν ε, δεν απαντήσω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση ε, παρακαλώ να επανέλθετε και αν μπορώ να επεκταθώ θα επεκταθώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την παρατήρηση του κυρίου Έλερ όσον αφορά τη υφιστάμενο δίκτυο δομών ε, κυβερνοασφάλειας που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, σύμφωνα με την ΕΝΗΣΑ, όπως αναφέρατε, σε κάθε χώρα έχουμε διάφορες ε, δομές ε, και μιλήσατε συγκεκριμένα για μία η οποία συντονίζει και πράγματι συντονίζει αυτό κάνει. Αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι λείπει θα ε, μπορέσουμε, ελπίζουμε να το βελτιώσουμε και θεωρούμε ότι είναι ακριβώ αυτό το νέο θέμα των αρμοδιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφαλείας γιατί πρέπει να δίνουμε ε, την πολιτική του να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Η τάση στον κόσμο της κυβερνοασφαλείας είναι η αμυντική μηχανισμοί. Συμβαίνει το συμβάν αλλά η ε, κακοήθης ε, πράξη πάντα έχει μεγάλη δημιουργικότητα. Οπότε είναι σημαντικό και εδώ πέρα έρχομαι στο ερώτημα του κυρίου Νίκας γιατί είναι σημαντικό να έχουμε αυτά τα κέντρα αριστείας κυβερνοασφάλειας γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο της έρευνας οπότε κάνουν την έρευνα και τελικά πηγαίνουμε προς ε, ένα ευρωπαϊκό κέντρο το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τα εθνικά κέντρα και θα μεταφραστούν τα ερευνητικά ευρήματα σε βέλτιστες πρακτικές για να διασφαλίσουμε τις δημοκρατικές μας αξίες και οι πολίτες ε, να έχουν εμπιστευτικότητα αλλά και ένα λογικό επίπεδο διαθεσιμότητας ε, των δεδομένων αυτών ε, στον κοινωνικό και στον εμπορικό τομέα. Οπότε να έχουμε κάποιες δομές συντονισμένες, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάποιες ε, περισσότερες προσπάθειες και βεβαίως να ρίξουμε και περισσότερο χρήμα στην πλευρά της έρευνας και να πάρουμε αυτό το έβριμα και να το βάλουμε στις βέλτιστες πρακτικές. Τώρα για την ερώτηση του κυρίου Νίκα, η παρατηρήσή σας είναι πολύ καλή. Όπως και η ερώτηση. Ένα τμήμα της απάντησης βρίσκεται στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Έλλερ. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην έρευνα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σήμερα ξέρετε ότι έχουμε και έναν οργανισμό αρμόδιο στη Ρουμανία, τον λεγόμενο CERT, που είναι ο κύριος παίκτη σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της κυβερνοασφάλειας στη Ρουμανία. και ε, θα ήταν πολύ καλά, καλό μέσα αυτών των νέων ε, κέντρων ε, να επικεντρωθούμε στην έρευνα και να μπορέσουμε να δώσουμε ένα βήμα προς τα μπρος για να μπορέσουμε να αποθήσουμε τις επιθέσεις σε ηλεκτρονικό επίπεδο. Τώρα, καθώς ε, μιλερουμενικά θα αναφερθώ και στι ερωτήσει του κυρίου Μαρινέσκου και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ό,τι δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Αναφερθήκατε σε ένα πρόγραμμα πλαίσιο. Αν κάνω λάθος να με διορθώσατε. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης. Ξέρω ότι εσείς ενεργοποιήσετε στο θέμα των μεταφορών. Το πρόγραμμα ο μηχανισμός συνδέοντα την Ευρώπη έχει τρεις σημαντικές συνιστώσει. Και πραγματικά δεν εκπλήσω μου θέσατε αυτή την ερώτηση, καθώ είναι η πιο σημαντική συνιστώσα σε ό,τι αφορά την κατανομή των κονδυλίων, ε, είναι οι μεταφορές. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ και αν μου επιτρέπετε στη ε, συγκεκριμένη δημοσιονομική κατανομή, γιατί στη συνέχεια αυτό εξαρτάται από συντονιστές και από τους ηγέτες που θα πάρουν τις αποφάσεις. Έχουμε τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά από τη δική μου άποψη υπάρχει, ε, είναι ένα πρόγραμμα που υπήρχε, ο Μηχανισμός Συνδέοντας στην Ευρώπη, και τώρα συζητάμε τον προϋπολογισμό για να συνεχιστεί από το 2021 μέχρι το 2027. Θα ήθελα να δω έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σύγκριση με το πρόγραμμα των προηγουμένων ετών, αλλά η μόνη δυνατότητα είναι να έχουμε ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές. Αν ισχύει αυτό και έχουμε ένα ξεκάθαρο φάκελο επενδύσεων, μπορούμε να ζητήσουμε και αυξημένους πόρους ανάλογα με τις φιλοδοξίες που θα προτείνουμε. Επίσης, εσείς αναφερθήκατε και σε άλλους διαδρόμους θα ήθελα όμω να επαναλάβω ότι είναι υπό συνεχή συζήτηση και διαπραγμάτευση ο φάκελο αυτός. Τα χρήματα που έχουμε σήμερα, τα κονδύλια για την ψηφιακή συνιστόσα του προγράμματος αυτού, σε μεγάλο βαθμό αφορούν επενδύσεις για τα ευρυζωνικά και την αύξηση του επίπεδου επικοινωνίας και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Θα προσπαθήσω να είμαι στον δυνατόν πιο γρήγορο. Ε, βλέπω ότι ο πρόεδρο μου κάνει νεύμα ότι θα πρέπει να βιαστώ. αναφερθώ λίγο στην ε, τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το οποίο είπε η κυρία Μιλνάρ και ο κύριος ε, να ανέφερε κάποια πράγματα και θα ήθελα κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε αυτά λεπτομερώς. Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ότι δεν είναι αρκετά παρούσα στο πρόγραμμα μας. Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και από την αρχή, βλέποντας διάφορους φακέλους, θεωρούσα ότι θα έπρεπε να έχουμε μια μεγαλύτερη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο. Γι' αυτό το πρώτο άτυπο σχετικό συμβούλιο που θα έχουμε τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την ψηφιακή ατζέντα στο Βουκουρέστι θα δείτε εκεί πέρα στην πρώτη σελίδα την τεχνητή νοημοσύνη. Προετοιμάζουμε το άτυπο συμβούλιο και θα έχουμε τελικά συμπεράσματα για το επίσημο συμβούλιο για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας ε, και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία ε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Συμφωνώ με αυτό το οποίο λέτε, ότι δεν το συζητάμε αρκετά, αλλά οπωσδήποτε θα έχουν ε, μεγάλη παρουσία αυτά τα ζητήματα. Επίσης, ε, κύριε Τσεζάκα, να πω δύο λόγια για την παρατήρησή σας σε σχέση με τα διάφορα κριτήρια για τους προμηθευτές για τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε και τι υπονοείτε και έχουμε ευτυχώς πολλούς και διάφορους προμηθευτές ε, της τεχνολογίας αυτής οπότε δεν βλέπω κάποιον λόγο ανησυχίας ε, όσον αφορά την εξέλιξη και το να περάσει η βιομηχανία στην πέμπτη γενιά. Δύο λόγια για την Ανατολική Γειτονία. Ε, πλησιάζουμε στην δέκατη επέτειο και ένα σημαντικό έγγραφο που είναι κομμάτι της διακήρυξης για την εναρμόνιση της ε, ψηφιακής αγοράς αφορά την εκπαίδευση και την έρευνα και τα αριθμιστικά ζητήματα για να έχουμε έτσι κάποιο κοινό του... Ναι, μπορώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Σύντομα όμως. Συντομεύεται. Λοιπόν, ο κύριος Ηλικιώτης. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα συνεχίσουμε τον ε, τριμερή διάλογο με την ψηφιακή Ευρώπη και σας διαβεβαιώ ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προχωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε όλους αυτούς τους ε, φακέλους. Κύριε Ζουρίνιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να είστε κάπως πιο συγκεκριμένος ε, για το τι εννοείται εισηγητής για την ψηφιακή οικονομία, αλλά μετά τις διευκρινήσεις που δώσατε μπορώ να σας πω ότι στο πρόγραμμα για την ε, ψηφιακή Ευρώπη έχουμε σήμερα μάλιστα τεχνικό τριμερή διάλογο, κάτι το είναι καλό σημάδι. Θα ήθελα να απαντήσω και άλλες ερωτήσεις, ε, αλλά ο χρόνος τελείωσε. Α, σύντομα, λέει ο πρόεδρος, αν μπορείτε πολύ σύντομα. Δεν ξέρω, απαντήθηκαν όλε. Νομίζω ναι, λέει ο κύριος Πετρέσκου. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό να ε, γίνονται τα ερωτήματα επισήμως στην συζήτησή μας ε, και ας μην απαντηθούν τώρα γιατί τα σημείωσε όλα η Ρουμανική Προεδρία ούτως ή άλλως. Και θα ήθελα τώρα να δώσω λόγο ξανά στον ε, κύριο Άντων, τον Υπουργό. Ευχαριστώ. Κύριε Έρνστ, ε, μία φράση θα σας πω. Ε, έχει μεγάλη σημασία να φροντίσουμε τις περιοχές που ζουν από τον άνθρακα γιατί σχεδόν όλοι όσοι έχουν αυτό το πρόβλημα έχουν το ίδιο πρόβλημα και το συζητάμε και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την πρωτοβουλία της Κομισιόν ε, για τις περιοχές αυτές αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να διευρυνθεί. Αυτά ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση. Ίσως ε, δεν υπήρχε αρκετός χρόνος ε, και σας ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι απαντήσεις, οι παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργή για την συνεργασία και φαντάζομαι τους επόμενους μήνες θα έχουμε συχνές συναντήσεις. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τη Ρουμανική Προεδρία. Πολύ σημαντικό. Σημαντική. Επίσης, έχουμε τον κύριο Νικολάε Χούντουκ, που είναι υπουργό Έρευνα και καινοτομία, Όχι μόνο έρευνα και καινοτομία, αλλά εν γέννη ατομική πυρηνική έρευνα, διάστημα, ίτερ, πολλά θέματα ό,τι σχετίζεται με την έρευνα, είναι στην αρμοδιότητά του. Και μετά έχουμε τον κύριο Νίκουλαε Μπανταλάου, που είναι Υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών, υπεύθυνο για βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία. Όλα πολύ ενδιαφέροντα. Minister, take Uh, Αγαπητοί μου φίλοι, στην αρχή θα έχουμε τον Υπουργό τον κύριο Νικολάη Ουρντουκ που ασχολείται με την έρευνα και την καινοτομία. Να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι έχουμε τον ορίζοντα Ευρώπη, το πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και καινοτομία συγκεκριμένο πρόγραμμα που εφαρμόζει, το, υλοποιεί το πρόγραμμα Horizon Europe, το διαστημικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Έρευνα και κατάρτιση, πρόγραμμα της ε, Ευρωπαϊκής ε, Εταιρείας Πυρηνικής Ενέργειας και σύμπραξη για το ΙΤΕΡ και ανάπτυξη της ενέργειας μέσω σύνδεξης. Έχουμε αρκετά θέματα προς συζήτηση στην περίπτωση της βιομηχανίας, πολύ σημαντικό αυτό, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που τελεί υπό διαπραγμάτευση και σαν πρόταση μη νομοθετικών νομοθετικού περιεχομένου, συντονισμένο πρόγραμμα για τεχνητή νοημοσύνη και ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική. Δεν είναι νομοθετικού περιεχομένου, αλλά είναι πολύ σημαντικά θέματα για τους πολίτες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεκινήσει λοιπόν η συζήτησή μας. Ζητώ συγγνώμη και από τους δύο υπουργούς που καθυστερήσαμε περισσότερο από το αναμενόμενο. Με ένα τέταρτο καθυστέρηση ξεκινάει η συζήτηση, αλλά νομίζω ότι έχουμε επαρκή χρόνο για μια ενδελεχή συζήτηση. Παρακαλώ τον Υπουργό Νικολάη Χουντούκ να ξεκινήσει την ε, συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε Μπούζεκ, Κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της ε, Ρουμανικής Προεδρίας για τον τομέα της έρευνας, της καινοτομία ε, και του διαστήματος. Όπως ε, όλοι γνωρίζουμε, η έρευνα αποτελεί έναν κινητήρα της ε, ανάπτυξης, μια μηχανή της ανάπτυξης όλων των κρετών. Και είμαι σίγουρος ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τομέας ε, της έρευνας θα είναι η κύρια μηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και θα έχουμε και αύξηση της ευημερίας όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να παραμπίνει ο κεντρικός κινητήρας πρόθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτή την έννοια θέλω να διευκρινίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και τις απαραίτητες υποδομές για να διατηρήσει μια ηγετική θέση σε ό,τι αφορά τον τομέα της επιστημονικής έρευνας. Και στο πλαίσιο αυτό, ο πιο σημαντικός φάκελος που συζητάμε στον τομέα της έρευνας είναι αναφεσβήτητα το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Ένα πρόγραμμα το οποίο ορίζει το θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, και την έρευνα από τον Ευρωπαϊκό, που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Στην δική μας ε, συζήτηση, στην ε, συζήτηση του Συμβούλου Ανταγωνισμού, στο Συμβούλιο έχουμε 7 φακέλους, οι 6 αφορούν τον τομέα της έρευνας και ο ένας φάκελος στο διάστημα. Στον τομέα της έρευνας, Όπως είπα, ο πιο σημαντικός φάκελος είναι ορίζον Ευρώπη. Υποτελείται από δύο συνιστώσεις, το πρόγραμμα πλαίσιο και τα συγκεκριμένα προγράμματα. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο, θέλω να υπογραμμίσω ότι η Αυστριακή Προεδρία κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την επιτάχυνση των συζητήσεων. Έτσι, Μόνο 7 μήνε από την έναρξη των εργασιών επί του φακέλου αυτού κατορθήσαμε να φτάσουμε σε τριμερεί διαλόγου ε, στι αρχέ Ιανουαρίου. Στι 9 Ιανουαρίου είχαμε τον πρώτο τριμερή διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβουλίου. Εμεί αναλαμβάνουμε τη δέσμευση, να καταβάλουμε τι ίδιε προσπάθειε σε ό,τι αφορά την ε, ταχύτητα πρόθεση αυτού του φακέλου έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη το 2021. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ειδικά προγράμματα, μπορούμε να αναφέρουμε το εξής. Είναι ένα βήμα πίσω, γιατί συνδέονται άμεσα με το πρόγραμμα πλαίσιο ιδανικά θα ήταν ε, καλό να μπορέσουμε να έχουμε μια γενική μερική συμφωνία μέχρι το τέλος της Ρουμανικής Προεδρίας. Ακολουθούν άλλοι δύο φάκελοι που συνδέονται με το Horizon Ευρώπη. Ο φάκελος ε, European Open Science Cloud και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Κοινοτομίας. Αυτοί οι δύο φάκελοι δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Άρχισαν οι συζητήσεις ε, στα μέσα του 2018, όμως είναι και θα γίνουν δύο βασικοί πυλώνε του προγράμματος Horizon Ευρώπη. Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Νέφος της Ανοιχτής Επιστήμης, Open Science Cloud, εισάγει μια νέα ενία ανοιχτής επιστήμης και θα επιτρέψει πρόσβαση στα αποτελέσματα των ερευνών ε, τόσο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και στις επιχειρήσεις αλλά και σε όσους εργάζονται στην ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε στην εθνική νομοθεσία ταχύτερα τα αποτελέσματα της έρευνας που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καιροτομίας και Τεχνολογίας, εδώ η Κομισιόν έχει προτείνει κάποιες τροπολογίες στον κανονισμό προκειμένου το Ινστιτούτο να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικό στην εφαρμογή των στόχων του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη. Και πάλι, στον τομέα της έρευνας έχουμε δύο ακόμη πιο ευαίσθητους φακέλους. Μιλάμε για το Euratom. Ξέρουμε ότι ένα μέρος των κρατών μελών έχουν κάποιους δισταγμούς σε σχέση με τη χρήση της πυρηνικής και θα ήθελα να υπογραμμίσω πως όταν συζητάμε για έρευνα στα πυρηνικά, δεν θα πρέπει απαραίτητα να σκεφτόμαστε μόνο την πυρηνική ενέργεια, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τους συναφείς τομείς όπου έχουμε πυρηνική έρευνα, όπως παραδείγματο χάρη στην ιατρική. Και θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, η θεραπεία του καρκίνου. δεύτερο φάκελο, το ΤΕΑΠ. Αυτοί οι δύο φάκελοι ε, παρουσιάστηκαν στην προσοχή της Επιτροπής το του 2018. Έτσι λοιπόν ε, θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τις συζητήσεις. έτσι ώστε ιδανικά αν ευνοήσουν οι συνθήκες να έχουμε μια γενική μερική συμφωνία μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Και τέλος ο τελευταίος φάκελος που έχουμε στη συζήτηση αναφέρεται στο διάστημα. σε αυτό το φάκελο και πάλι μπορούμε να προτείνουμε την επίτευξη Γενικής Μερικής Συμφωνίας, μια PGA, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Πρόκειται για μια σειρά προγραμμάτων για το διάστημα που υλοποιούνται τη στιγμή αυτή και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τον Γαλιλαίο, τον Κοπέρνικους, το Έγνος. Πρόκειται για προγράμματα που δίνουν ε, στοιχεία σε σχέση με την τοποθεσία πληροφορίες σε επίπεδο χώρου. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η δική μας άποψη θα ήταν ότι αυτά τα προγράμματα είναι μη στρατιωτικού χαρακτήρα και θα πρέπει να παραμείνουν τέτοια. Σας ευχαριστώ. Προσπάθησα να σεβαστώ τα 7 λεπτά, αλλά ξεπέρασα το χρόνο κατά 2 λεπτά. Ελπίζω να μην είναι μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπουργέ, για την παρουσίασή σας, την ομιλία αυτή. Τώρα, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο ε, Μπανταλάου. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Έχω την τιμή να βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σα για να παρουσιάσω τι προτεραιότητε και τι κύριε πτυχέ τη προεδρία τη Ρουμανία στο Συμβουλίο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στον τομέα τη αρμοδιότητά μου, δηλαδή ανταγωνιστικότητα και βιομηχανία. Ένα τομέα ε, που εντάστηκε στι αρμοδιότητε τη επιτροπή Ήτρα. Καταρχήν θέλω να επαγραμμίσω το γεγονό ότι η Προεδρία τη Ρουμανία αποτελεί μια καθοριστική Προεδρία σε ό,τι αφορά την εντολή, τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη στο να διαχειριστούμε την νομοθετική διαδικασία. Γι' αυτό οι προσπαθίες μας επικεντρώνονται στο να προχωρήσουμε στους νομοθετικούς φακέλους όσο το περισσότερο δυνατόν τους πρώτους τρεις μήνες του έτους. Οι προτεραιότητες της Προεδρίας μας στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανίας στοχεύουν στη βιομηχανική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ψηφιοποίηση και την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα επίκαιρα στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο και είναι πάρα πολύ σχετικά στο σημερινό κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Η προσαρμογή των βιομηχανικών οικοσυστημάτων στην ψηφιοποίηση αποτελεί μία πρόκληση και μπορεί να μεταφορθεί σε ευκαιρία για την αύξηση της ε, βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης την επόμενη δεκαετία. Η ψηφιακή μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν τους κύριους παράγοντες που θα συνεισφέρουν ε, στην χάραξη της βιομηχανικής πολιτικής ε, του 2030 γιατί θα είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε κατάλληλες ικανότητες. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο «Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη και το σχετικό παράρτημα» προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο την πρόθεση της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και εκτιμάμε το γεγονό ότι αυτή η κοινοποίηση της Επιτροπής βασίζεται στις ακόλουθες ιδέες, κοινά σχέδια και συμπληρωματικές προσπάθειες, ανάπτυξη της ΔΙΤ και μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τις νοσίστατες επιχειρήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ενδυνάμωση της ε, αριστείας ε, σε τεχνολογία ε, τεχνητής νοημοσύνης και η διάδοσή τους, η προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης για να προετοιμάσουμε την κοινωνία μας καλύτερα για την τεχνητή νοημοσύνη είναι δημιουργία ενός ε, χώρου ευρωπαϊκών δεδομένων ε, για την τεχνητή νοημοσύνη και για το δημόσιο τομέα. ανάπτυξη κωδικών ηθικής ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και να διασφαλίσουμε ένα ανοιχτό νομοθετικό πλαίσιο για την καινοτομία. Πτυχέ που συνδέονται με την ασφάλεια των εφαρμογών τεχνητή νοημοσύνη και υποδομέ για την διεθνή ασφάλεια η ανακοίνωση μας ε, δείχνει το γεγονός ότι ε, έχει δοθεί προτεραιότητα σε τομείς όπως είναι οι μεταφορές, η κινητικότητα, η ιατρική βοήθεια, η ασφάλεια και η ενέργεια για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Εκτιμούμε το γεγονός ότι το προσάρτημα στο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη ε, αναφέρει με τίτλο «Ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης Made in Europe 2018» κάτι που δείχνει την επιθυμία η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της, της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δράσεις που θα ξεκινήσουν φέτος ε, ή του χρόνου θα δημιουργήσουν δραστηριότητες ε, που θα υλοποιήσουμε και τα επόμενα έτη. Μεταξύ αυτών είναι και η πρόθεση των κρατών μελών να θετήσουν εθνικέ στρατηγικέ και να καθορίσουν προπολογισμού στα μέσα του 2019. Η Προεδρία της Ρουμανίας στο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει ένα σύνολο συμπρασμάτων του Συμβουλίου βάσει του σχεδίου δράσης για την τεχνητή νοημοσύνη που θα υιοθετηθούν στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 18 Φεβρουαρίου 2019. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι πτυχές που αναφέρονται στην τεχνητή νοημοσύνη θα συζητηθούν ε, σε ε, διάφορες συνεδριάσεις του Συμβουλίου λόγω του αντίκτυπου που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία τα επόμενα έτη. Κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής ε, Προεδρίας, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη βιομηχανία, ε, στην, ε, στα κλάστερ ε, και στις αλυσίδες αξίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική που να προσανατολίζεται στο μέλλον, ικανή να απαντήσει στις σημερινές προκλήσεις. Αυτή η πτυχή αναδείχθηκε και στην δήλωση των Παρισίων στις 18 Δεκεμβρίου 2018 από 18 κράτη-μέλη κατά την έκτη διάσκεψη φίλη της βιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, όπου ανήκουν και μικρές και μισές επιχειρήσεις, χρειάζεται μία μικροπρόθεσμη πολιτική με ένα όραμα τουλάχιστον μέχρι το έτος 2030 που να λαμβάνει υπόψη την επικοινομορφία της σημερινής βιομηχανικής βάσης ε, και να ε, μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δίνονται από την ψηφιοποίηση, την καινοτομία, την κυκλική οικονομία και την απαρθρακοποίηση τομείς που, καθορίζονται, θα καθορίσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η διατήρηση μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να διασφαλίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία ε, και ε, σημαντικό βάρος προϊόντων με μεγάλη προσθέμενη αξία στις εξαγωγές είναι ουσιαστική για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό το όραμα βρίσκεται στο δικό μας ευρωπαϊκό θεματολόγιο και ισχύει και για τη Ρουμανία όπου το βάρος της βιομηχανίας στο ΕΠ είναι πάνω από 25%. Κατά την άποψή μας ε, χρειάζεται και προστασία της ανταγωνιστικότητας ε, των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τη συστηματική ένταξη της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης και θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε συζητήσεις ε, τόσο για τους παράγοντες που επηρεάζουν την μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, αλλά και σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή. Η πραγματικότητα σήμερα μας δείχνει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα χωρίς ψηφιοποίηση, χωρίς τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Ο δικός μας κόσμος και ο κόσμος των παιδιών μας ε, γίνεται όλο ένα και πιο ψηφιακός και η στενή σχέση μεταξύ της έβρεσης θέσης εργασίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι περισσότερο προφανής παραποτέ. Ε, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Προς αυτό το σκοπό, οι επενδύσεις στην υποδομή, της ψηφιακές ικανότητες και την κοινοτομία αποτελούν υποχρεωτική συνθήκη. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία της ψηφιοποίησης των εταιριών αυξάνεται γιατί αυτές συνειδητοποιούν το δυναμικό που προτείνουν οι ψηφιακές λύσεις ε, και ε, ότι αλλάζουν οι προσδοκίες των καταναλωτών. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, ε, Έχουμε κάποιες εταιρείες που απέκτησαν πολύ μεγάλη αξία και δραστηριοποιούνται σε τομείς πληροφορικής και επιγραμμικού εμπορίου. Η Προεδρία θα προτείνει ένα σύνολο συμπρασμάτων του Συμβουλίου για το θέμα της βιομηχανίας, που θα παρουσιαστεί στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27 Μαΐου 2019. Αυτά θα περιλαμβάνουν ε, και τα αποτελέσματα των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα στην ε, διάσκεψη ημέρες Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας 2019 και σε άλλα φόρα αλλά θα συμπεριλάβουμε και τις απόψεις της βιομηχανίας. Ελπίζουμε ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα προσανατολίσουν την επόμενη Επιτροπή να παρουσιάσει μία θεματική ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιστική από τη σκοπιά της βιομηχανίας που να περιλαμβάνει και αναφορές στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Όπως ε, γνωρίζετε, η Γενική Αμερική Συμφωνία ε, επιτεύχθη υπό την Αυστριακή Προεδρία και είχαμε τον πρώτο τριμερή διάλογο 16 Ιανουαρίου. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε βάσει της πρόσφατης συμφωνίας μας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ε, Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας να συνεχίσουμε να δασιζόμαστε σε αυτό. Σας ευχαριστώ και ε, θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα θέματα όπως πρέπει στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Τώρα, να ξεκινήσει η συζήτησή μας με τους ε, συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Έλερ είναι πρώτος από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ήδη από την Αυστριακή Προεδρία, οι δύο εισηγητέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Ορίζοντα Ευρώπη είπαν ξεκάθαρα στους 28 υπουργούς, του αρμόδιους για την έρευνα, πως το περιεχόμενο και η έγκαιρη έναρξη θα πρέπει να επικρατήσει των εσωτερικών διαφωνιών των Υπουργών. Οπότε έγινε μια εξαιρετική προσφορά προς το Συμβούλιο να μην υπάρχει διπλή νομική βάση του προγράμματος προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Καινοτομία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2020 αν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες για τις εκπομπέ και μετά να αρχίσουμε ε, την ε, κατάρτιση των προγραμμάτων του 2020. Ο πρόεδρος Μακρόν, οι αρχηγοί των κρατών ε, αποφάσιζαν ε, για μια καινοτόμο Ευρώπη και αυτό κάνουμε κι εμείς. Υπό τον όρο λοιπόν ότι θα μπορέσει να αντισταθμίσει κάπως το δικαίωμα της συναπόφασης και το δικαίωμα της εξέτασης το Συμβούλιο, ελπίζουμε πριν το τέλος της θητείας. Όσον αφορά δε τα συγκεκριμένα προγράμματα, ε, θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να διατηρηθεί η πρακτική του προγράμματος πλαισίου 7, δηλαδή να επιτύχουμε μια πολιτική συμφωνία και για την συναπόφαση και για την διαβούλευση για τα πακέτα τα οποία είναι νέα προγράμματα πλαίσιο. Οπότε ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να δοθεί μια σαφής διαπραγματευτική εντολή στην Προεδρία ανεξαρτήτως ε, επίπεδου και μορφής, αλλά πριν το τέλος του Φεβρουαρίου 2019. Με το να μην κάνουν κάτι τέτοιο, προφανώς ε, το Συμβούλιο θα καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα πριν από το τέλος της θητείας. Πέρα από κάποιες αρνητικές εξωτερικότητες, οι συζητητέ θέλουν να τονίσουν πως το Συμβούλιο θα χάσει ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρία για να λύσει γρήγορα το θέμα της νομικής βάσης και να προλάβει την συνέχεια των περαιτέρω πολιτικών διαπραγματεύσεων. Οπότε ζητάμε πραγματικά από την Προεδρία να καταλήξει σε μια συμφωνία στο Συμβούλιο, μια συμφωνία επί της αρχής ε, για το πρόγραμμα στο σύνολό του, γιατί για να διαβεβαιώσουμε τους Ευρωπαίους ερευνητές ε, ότι έχουμε μια ατζέντα καινοτομία, έχουμε οικονομικό ζήτημα, έχουμε τον κοινωνικό τίτλο και οι πολίτε τη Ευρώπη αναμένουν να κάνουμε κάτι. Uh, thank you very much, Uh... Σας ευχαριστώ. Ισχυρό το μήνυμα. Όταν έχετε ένα μήνυμα βεβαίω πάντα είναι δυνατό. Ο συναδελφό Νταν Νίκα. Ευχαριστώ. Θέλω να χαιρετήσω τους δύο υπουργού και να τους πω ότι οι προσδοκίε από την πλευρά του Κοινοβουλίου είναι πολύ μεγάλε. Έχουν ε, στη διάθεσή του μόνο 3,5 μήνες και όχι μόνο έξι μήνε. Οι φάκελοι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι. Και ταυτόχρονα να σα πω ότι αυτή η Επιτροπή ασχολείται με το 80% των θεμάτων της οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ασχολούμαστε με γεωργία και βιομηχανία. Κατά τα υπόλοιπα, όλη η έρευνα και η βιομηχανία είναι αρμοδιότητα αυτή τη Επιτροπή. Ε, θα ήθελα να περάσω σε ένα σημαντικό θέμα. Είμαι συντονιστή, ε, συγγνώμη, είμαι για το Horizon Europe και νομίζω το μήνυμα του κυρίου Χορντούκ πρέπει να το διαβάσετε στο Συμβούλιο. Εδώ έχουμε τους εισηγητές ε, και τους κοιόδης εισηγητές και είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοθέτημα αναφέρομαι και στο πρόγραμμα πλαίσιο αλλά και στα συγκεκριμένα προγράμματα. Είχαμε ανοιχτό πνεύμα, ήρθαμε με μεγάλη εμπιστοσύνη στον πρώτο τριμήρη διάλογο, αλλά δυστυχώς ε, φαίνεται ότι από την πλευρά του Συμβουλίου δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας. Και αυτό θα ήταν μεγάλο χτύπημα για όλη την ε, ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, γιατί χρειάζεται χρόνος να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει το 2021 και δεν ε, νομίζω ότι πρέπει εδώ να παίζονται παιχνίδια. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Ξέρουμε ότι η Ρουμανική Προεδρία δεν ε, μπορεί να επιβάλλει κάτι στο Συμβούλιο, αλλά πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι φτάνει πια. Είναι άθη συνάθλη ο μιλητή στα αγγλικά. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια είναι τα στοιχεία διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, δεν ε, θα χάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ε, ετοιμάσαμε την έκθεση μέσα σε 6 μήνες, κάναμε κάθε προσπάθεια για να προετοιμάσουμε και να είμαστε εντελώ ανοιχτοί, αλλά τελικά αν θα χάσουμε, επειδή το Συμβούλιο θα βρει κάποια επιχειρήματα και κάποιες δικαιολογίες, αυτό δεν θα το ανεκτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, ομόφωνα σας το λέμε αυτό. Δηλαδή ε, παρακαλώ να διαβιβάσετε αυτό το μήνυμα από μας ξεκάθαρα και ελπίζουμε στον επόμενο τριμερή διάλογο να δούμε ποια είναι η απάντηση του Συμβουλίου και φυσικά ε, επιφυλασσόμαστε για τις συνέπειες. Κύριε Υπουργέ Μπαντελάου, μιλήσατε για κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μας, για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπατε ότι αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων παγκοσμίω. μπορείτε να μα πείτε περισσότερε λεπτομέρειε για το θέμα αυτό, γιατί είχε συνεχή ανησυχία το Κοινοβούλιο σε σχέση με το πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα τη τεχνητή νοημοσύνη γιατί θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια μεγάλη και σημαντική δύναμη στον κόσμο και η τεχνητή νοημοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο. Έχουμε βέβαια και άλλα προγράμματα παράλληλα. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για να μπορέσετε να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα από τα οποία εξαρτάται η ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκ μέρους του ECR. Για το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Εγώ ήθελα τον λόγο για το επόμενο θέμα που ε, ασχολεί, απασχολεί τον κύριο Τουσανόφσκι για το Ταμείο Άμυνας ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να ρωτήσω τώρα, ε, είναι το ίδιο θέμα? Λοιπόν, Προσεχώς ε, θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δύσκολες διαπραγματεύσεις μας ε, και θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπει η Προεδρία τις πιθανότητες ε, να τα καταφέρουμε μέχρι τις ευρωεκλογές αρχές Φεβρουαρίου ουσιαστικά να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Άκουσα μόνο τα τελευταία λόγια του κυρίου Υπουργού είπε το πόσο σημαντικό είναι να συνεισφέρουμε στην ε, εξέλιξη της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας και νομίζω ότι θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο να συνεισφέρει σε αυτό ως ε, μια όθηση στην καινοτομία Και καλό θα ήταν, δεν είναι τόσο τεράστιο το χάσμα, να ολοκληρωθούν αυτά τα ζητήματα μέχρι τις ε, ευρωεκλογέ. Θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να κάνετε εξ ονόματος ε, Προεδρίας και Συμβουλίου μία δήλωση προθέσεων. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βίρινγκ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Ουρντουκ, ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Η ερώτησή μου σχετίζεται με την ερώτηση του κυρίου Νίκα και του κυρίου Έλερ. Η Ρουμανική Προεδρία τι θα κάνει να εξασφαλίσει έγκαιρη έναρξη του νέου προγράμματος πλαισίου. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου. Το περιεχόμενο και η έγκαιρη έναρξη θα πρέπει να επικρατούν έναντι διοργανικών διαμαχών για τη νομική βάση του προγράμματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλίνη. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καλή εντολή για διαπραγματεύσει για το διάστημα πλευράς Ευρωκοινοβουλίου. Η εντολή σας δεν είναι τόσο πλήρης. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Πότε θα γίνουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά το συνολικό κείμενο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαστήματος. Δεύτερη ερώτηση. Στην εντολή μας έχουμε σαφή εντολή για πυλώνες. Θέλουμε τον κατάντη τομέα διακυβέρνηση, σωστή διακυβέρνηση, χωρίς επικαλύψεις και θέλουμε αυτόνομη πρόσβαση ε, στο διάστημα. Αυτός είναι πραγματικός πυλώνας για μας. Οι δικές σας προτεραιότητες για το διάστημα ποιες είναι. Τρίτο, νέο προγράμματα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη συνέχεια για τα προγράμματα πρώτης γραμμής. Γαλιλαίος, ε, Κοπέρνικος, Έγνος, πρέπει να βελτιώσουμε και νέα προγράμματα για να είμαστε ασφαλεί, Όπω το SSA και το GovSat.com. Ποια είναι η άποψή σα για τα νέα προγράμματα. Τέλο, είσαστε και υπουργό Έρευνα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια είναι η άποψή σα για τη συνεργασία μεταξύ του Horizon Europe και του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματο. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Ζωρίνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα κλειδί που τίθεται εδώ στη Ρουμανική Προεδρία συμπίπτει με το τέλος της θητείας και με τις ευρωεκλογέ. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία επί της αρχής για τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2020. Νομίζω ότι να έχουμε περισσότερε φιλοδοξίε είναι ουτοπικό. Όμω θα μπορούσαμε να έχουμε μια συμφωνία από τι αρχέ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα με τους υπόλοιπους φακέλους με ολοκληρωμένο τρόπο για το τον ορίζοντα, για το φάκελο για το διάστημα, για την ψηφιακή Ευρώπη, για την κοινή άμυνα προκειμένου σε αυτό το στάδιο, καθώς προσεγγίζουμε τις εκλογές, να ενισχυθεί η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, η ανταγωνιστικότητά μας και είναι πολύ σημαντικό με αυτά τα μικρά αποτελέσματα να τα κοινοποιεί η Ρουμανική Προεδρία. Γιατί, ξέρετε, ε, μετά τις εκλογές ε, να μην βρεθούμε στο μηδέν, δηλαδή να έχετε μία φιλόδοξη Προεδρία και που θα αφήσει το αποτύπημά της ε, και να μην επιτρέψει να κυρωθούν τα αποτελέσματα λόγω των εκλογών. Ευχαριστώ κύριο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου ε, του κύριου Κάριν, ο οποίο είναι συντονιστή του ΕΛΚ. Γιατί μόλι εξελέγει η πρωθυπουργό στη Λετωνία και γι' αυτό δεν ε, βρίσκεται εδώ. Είναι ο συντονιστή του ΕΛΚ, ο ε, κ. Κάριν, συντονιστή του ΕΛΚ για αυτή την επιτροπή. Έχω κάποιε ερωτήσει το ITER είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα σύντηξης, διαφορετικό από την πυρηνική ενέργεια. Δυστυχώς το Συμβούλιο όμως αποφάσισε να μην έχουμε διαδικασία σε συναπόφαση για το φάκελο αυτό. Υπάρχει δέση φυσικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι για εσάς δεν θα είναι ιδιαίτερα πολύ να, κάνετε μια, να έχετε μια μερική συμφωνία. Γιατί φυσικά δεν προβλέπονται τα κονδύλια. πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους, όπως είδατε. Κατά την άποψή μου, έχετε μια πολύ σημαντική αποστολή. Να διασφαλίσετε ίσες ε, συνθήκες για όλους τους ερευνητές και ιδίως για τους νέους, αλλά και για όσους προέρχονται από χώρες που δεν είχαν ακόμη πρόσβαση στα ερευνητικά προγράμματα, γιατί το πρώτο κριτήριο είναι η οριστεία και δυστυχώς ε, δεν κατορθώσαμε να βάλουμε ορισμό της αριστείας στο φάκελο που να διασφαλίζει τις ευκαιρίες για όλους. Θα σας παρακολούσω επίσης και εξ του κυρίου Σελήνη στο πρόγραμμα για το διάστημα να εξασφαλίσετε τον προπολογισμό για το έγκνος για να καλυφθεί όλη η Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ρουμανία δεν καλύπτεται στο σύνολό της για τον κύριο Μπεντελάου. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σκέφτεστε να διασφαλίσετε μια γεωγραφική ισορροπία στο πρόγραμμα άμυνας, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ στο Κοινοβούλιο, καθώς ε, πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα τέτοιου τύπου και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, αναφερθήκατε στην βιομηχανική πολιτική. Μπορείτε να μου πείτε ποιες συγκεκριμένε προτάσεις έχει η Ρουμανική Προεδρία στο θέμα αυτό, συγκεκριμένες όμως, προκειμένου να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική στο πιο ψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Okay. Uh, Καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερώτηση, απευθυνόμενη και προς τους δύο υπουργούς. Θα μπορούσατε να απαντήσετε σε ερωτήσεις και να προβείτε στα τελικά σας σχόλια, αν έχει την καλοσύνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω με το πιο καυτό θέμα, το πιο κανθόδες, που σχετίζεται με το πώς προχωρούν οι συζητήσεις για το πρόγραμμα πλαίσιο. Υποψιάζομαι ότι ο κύριος Έλλερ θα ήθελε να ακούσει μια απάντηση για τα ειδικά προγράμματα να διευκρινίσω εδώ ότι δεν μπορώ να πω την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να εκφράσω την άποψη του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο θέμα αυτό. Θέλω να σας πω όμως ότι τα ειδικά προγράμματα σχετίζονται πάρα πολύ στενά με το πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε το διάλογο που ξεκίνησε ήδη και λαμβάνονται σημειώσεις και σημειώνονται οι απόψεις ε, των ε, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στους τριμερείς διαλόγους που σχετίζονται με το πρόγραμμα πλαίσιο. Υπάρχει λοιπόν ένα συσχετισμός και τελικά τα δύο αυτά προγράμματα είναι ε, πολύ στενά συνδεδεμένα και τα ειδικά προγράμματα δεν μπορούν να βγουν από τις παραμέτρους του προγράμματος πλαισίου. Ίσως θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο και να προσπαθήσουμε να εργαστούμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να υπάρξει μια νέα απόφαση. Άλλωστε, το Φεβρουάριο έχουμε Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα. Εγώ από τη δική μου σκοπιά θα προσπαθήσω να μάθω ποια είναι η άποψη των συναδέλφων. Θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε και να δούμε πώς ε, μπορούμε να επιταχύνουμε την εξέλιξη των φακέλων. Δυστυχώς έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τις ε, ευρωεκλογέ. Από διοικητική σκοπιά μας συντομεύουν τη θητεία. Όμως, όπως σας είπα, όλα εξαρτώνται από την απόφαση του Συμβουλίου. Να προσπαθήσουμε να μετακινήσουμε τα πράγματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το διαστημικό πρόγραμμα, να σας πω ότι αύριο θα έχουμε συνάντηση με την Ερμόδια Επίτροπο και θα συζητήσουμε τη στρατηγική προσέγγιση, να δούμε ποιε είναι οι προτάσει της Κομισιόν για το διαστημικό πρόγραμμα. Όπως ξέρετε, Υπάρχουν δυνατότητες να ενταχθούν ορισμένες συνιστώσεις ε, του διαστημικού προγράμματος στο Horizon Europe. Σε σχέση τώρα με τον ορισμό της αριστείας, αν κατάλαβα καλά. Σίγουρα. Υπάρχουν ε, κλασικά συστήματα που μας επιτρέπουν να ιεραρχήσουμε τα μενεπιστήμια, τα ιδρύματα, τους ανθρώπους που υλοποιούν ερευνητικέ δραστηριότητες. Και σίγουρα υπάρχουν ε, διάφορες μέθοδοι, υπάρχουν και κριτικές ε, σε ό,τι αφορά αυτές τις αρχές. Ε, για το πώς μετράμε την αριστεία Βέβαια, εδώ μπορεί να ήταν ενδιαφέρον να εφαρμοστούν κάποια συστήματα αξιολόγησης ε, blind, blind μάλλον εννοεί ο μιλητής τυφλά συστήματα, δηλαδή να μην ε, γνωρίζουμε τα άτομα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Τώρα, να πάμε στο θέμα της βιομηχανίας και της αμυντικής βιομηχανίας. Έχετε το λόγο, Υπουργέ Μπεντελάου. Giving the last remarks. Για να απαντήσετε τι ερωτήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σε σχέση με όσο είπε ο κύριο Ντανίκα. Όταν αναφερθήκατε στους 3,5 μήνε, ήσασταν ε, πολύ αισιόδοξο. Μάλλον πρέπει να βιαστούμε πολύ περισσότερο, γιατί θα είναι πολύ πιο σύντομη η περίοδος για να μπορέσουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Να σας απαντήσω στην ερώτησή σας. Να σας πω ότι σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία εντός του Συμβουλίου. Το σχέδιο εκπονήθηκε βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής και του Σχεδίου Δράσης που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2017. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται και οι προηγούμενες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας και θέλω να σας πω ότι έγινε πολύ μεγάλη πρόοδος κατά την περίοδο της Αυστριακής Προεδρίας σε αυτό το τομέα. Τα συμπεράσματα μας δείχνουν τη σημασία που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μέσω ε, χωρών που θέλουν να αφιερωθούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, φαίνεται η σημασία των συνεργειών μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των βιομηχανικών τομέων. Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας όπου προσεγγίζεται και η σημασία της ε, κατάρτισης των επαγγελματιών για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και των μηχανικών καθώς ε, και πρέπει να στοχεύσουμε στις επιστήμες, στη μηχανική και στα μαθηματικά. Επίσης αναφέρεται και η εφαρμογή κώδικα δεντολογίας ε, που δημοσιεύτηκε ως σχέδιο στην ομάδα υψηλού επίπεδου για την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά τα συμπεράσματα τα έχουμε και προτείνουμε να υιοθετηθούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Φεβρουαρίου 2019. Σας ευχαριστώ. Pentru domnul profesor. για τον καθηγητή Κρασνοτεύσκη. Καλά το πρόφερα το όνομά σα. Να σας πω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο το υλικό, αλλά μας πίεζε ο χρόνος και προσπάθησα να είμαι σύντομος. Όπως είδατε και εσείς ότι το Ταμείο Άμυνας είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το νομοθετικό φάκελο για το Ταμείο Άμυνα. να σας απαντήσω για το ποια είναι η προσέγγισή μα. Η Γενική Αμερική Προσέγγιση επιτεύχθηκε υπό την Αστρική Προεδρία. Ήδη είχαμε τον πρώτο τριμερή διάλογο στι 16 Ιανουαρίου. Χαιρόμαστε που λαμβάνουμε διασφαλίσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη διαθεσιμότητα να κλείσουν οι διαπραγματεύσει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Αυτή την οδό θα θέλαμε να ακολουθήσουμε και ευχαριστούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δεσμευσή αυτή. Για αυτό τον τόσο σημαντικό φάκελο. Η ταχύτητα της ε, ανάλυσης του φακέλου αυτού σέβεται τη φιλοδοξία όλων. Όπως ξέρετε, η δική μας σκοπιά φαίνεται να έχει πολλά κοινά με τη δική σας, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να εντοπίσουμε μια συμβιβαστική λύση που να απαντά στις δικές μας ανησυχίες και να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που να λειτουργεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε βάσει της ε, συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Τομέα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από αυτού. Θα ήθελα να απαντήσω και στον κύριο Μαρονέσκο. Έθεσε μια αρκετά δύσκολη ερώτηση σε σχέση με τη γεωγραφική ισορροπία ή πώς αυτό θα επηρεάσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Θα ήθελα να σας απαντήσω στην ερώτηση αυτή, Όμω, ε, υπάρχει μια διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί με αυτό το ταμείο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο που να καλύπτει όλα τα κρατημέλη, την έρευνα κτλ. Όμω, ε, υπάρχουν τώρα διαπραγματεύσει μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τι ικανότητέ του και με τη γεωγραφική κάλυψη. Ανάλογα και με τους κινδύνους που βρίσκονται στην ε, εγκύτητά τους. Ξέρετε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό και από άλλη σκοπιά για το θέμα της γεωγραφικής ε, κατανομής. Όμως, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν συμπράξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να τις αναπτύξουμε για το Ταμείο Άμυνας. Για τον κύριο Μαρινέσκο και πάλι για το θέμα της βιομηχανίας, της βιομηχανικής στρατηγικής. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια η πολιτική της Κομισιόν ε, ήταν ε, η βιομηχανία, η βιομηχανική στρατηγική να χαράζεται ανάλογα με την κάθε ζώνη. Όταν μιλάμε για το περιβάλλον, το σκάρι, υπάρχει βούληση να έχουμε ένα ξεχωριστό τομέα με τον οποίο να συζητάμε για το θέμα της βιομηχανίας. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και θα έπρεπε να περιλαμβάνει οπωσδήποτε όλα τα κράτη-μέλη, ξεκινώντας από την παραγωγή της ενέργειας, μέχρι την παραγωγή αγαθών μεγαλύτερης προσθέμενης αξίας. Αν δεν σας ικανοποίησαμε την απάντησή μου, μπορείτε να μου πείτε να σας απαντήσω λεπτομερέστερα. Σας ευχαριστώ. Okay, uh, thank you very much. Uh... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας τώρα που είναι η αρχή της Ρουμανικής Προεδρίας. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, για τα σχόλιά σας. Ε, επίσημη εναρτήρια ε, τελετή για τη Ρουμανική ε, Προεδρία σήμερα στο Ευρωκοινοβουλίο, στο ίδιο κτίριο, στο ΖΑΝ, στον τρίτο όροφο, στις 18.30. Σε μία ώρα και 40 λεπτά. Σε μία ώρα και 40 λεπτά τρίτος όροφος, έναν όροφο πιο πάνω. Είμαστε στο δεύτερο όροφο. Επίσημη λοιπόν έναρξη, η τελετή της επίσημης έναρξης της Ρουμανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς και θα συνεργαστούμε τους επόμενους μήνες. Δίκιο έχετε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι το Φεβρουάριο. Τα πάντα είναι έτοιμα ακόμα και το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου ή δυνατόν. Έχουμε μερικές εβδομάδες μπροστά μας. Πολύ λίγες. Μπα τα καταφέρουμε όμως. Είμαστε προετοιμασμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί φίλοι, να σας χαιρετήσω. Thank you, Mr. Buzek. Thank you. Thank you very much. Dear φίλοι, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας ε, διάταξης. Ε, έκθεση για τις συνεχιζόμενες διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Το πρώτο θέμα είναι ο κύριος Σιλικιώτης. Η επανάχρηση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Έχετε πολύ καλά νέα κύριε Σιλικιώτη, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα είμαι αρκετά σύντομο. Ε, πρώτα απ' όλα, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και εισηγητές και τους συνεργάτες τους για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε αλλά και ιδιαίτερα στη γραμματεία τη ΙΝΤΡΕ για την υποστήριξη σε αυτή τη δουλειά. Πρέπει να πω δουλέψαμε συλλογικά ως ομάδα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτύχουμε τις βασικές προτεραιότητες που είχαμε θέσει εξ αρχής ως Κοινοβούλιο. Εν γέννη, πετύχαμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να διασφαλίζει πως η κοινωνία, οι πολίτες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι νέες αναδυόμενες επιχειρήσεις έχουν δωρεάν πρόσβαση σε πολύ σημαντικές πληροφορίες που κατέχει ο δημόσιος τομέας. Ειδικότερα, είχαμε επιτύχει να ενισχύσουμε τις αναφορές στην άγκη για προστασία των προσωπικών δεδομένων και να τονίζουμε την ανάγκη για πλήρη ευθυγράμμιση τη οδηγία PSI με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα. Πετύχαμε να διατηρήσουμε όλε τι εξαιρέσει που είχαμε ζητήσει για τι δημόσιε επιχειρήσει, διασφαλίζοντα έτσι το δίκαιο ανταγωνισμό σε σχέση με τι ιδιωτικέ επιχειρήσει που ακόμη δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία, ε, αναγνωρίζοντα και η Επιτροπή και το Συμβούλιο λογικό το επιχείρημα που πώ πρέπει να προηγηθεί ειδική έρευνα και εκτίμηση των επιπτώσεων ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε και τι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Δεχτήκαμε να διαγράψουμε την πρότασή μα από το άρθρο 1, αλλά με σχετική αναφορά στι ιδεολογικέ προτάσει, καλούμε τα κράτη-μέλη να μελετήσουν και να προχωρήσουν στην επέκταση τη οδηγία και στι ιδιωτικέ επιχειρήσει για να διασφαλιστεί έτσι δίκαιο ανταγωνισμό μέχρι να έρθει και η σχετική οδηγία από την Κομισιόν. Ενισχύσαμε στο κείμενο στο άρθρο 6 πω η πρόσβαση στι πληροφορίε πρέπει να είναι δωρεάν. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Πετύχαμε να γίνει αποδεκτή η λίστα που προτείναμε όσον αφορά τι κατηγορίε για βάσει των δεδομένων υψηλή αξία που θα δίνονται δωρεάν στην κοινωνία. Στη λίστα αυτή έχουμε βάλει πολύ σημαντικέ κατηγορίε βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων ε, και θεωρώ ότι αυτά αφορούν ε, ζητήματα που αφορούν και την καθημερινότητα του πολίτη αλλά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν ε, το περιβάλλον που σχετίζονται με εταιρείε και διασφαλίζουμε έτσι μεγαλύτερη επίσης διαφάνεια. Εξής σημαντικό είναι ότι ε, διασφαλίσαμε την εμπλοκή και την ενεργό μας δράση στην επιλογή των κατηγοριών και για το μέλλον μέσω της πράξης κατεξουδότησης του Τελεκεϊτάχτ η οποία απαιτείται για την επέκταση της λίστας. Πετύχαμε λοιπόν η λίστα να μπορεί να επεκταθεί μονάχα με την προσθήκη νέων κατηγοριών με κατεξουσιοδότηση πράξη, εφόσον βέβαια προηγηθεί επαρκή και ουσιαστική διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίση, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μειωθεί αυτή η λίστα με τι κατηγορίε όπω τι προτείναμε. Βεβαίω, τέλο, θέλω να σημειώσω ότι αποδεχτήκαμε ω συμβιβασμό και εμεί να δοθεί εκτελεστική πράξη, implementing act, όσον αφορά την εφαρμογή αυτών κατηγοριών και την επιλογή των συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων υψηλή αξία καθώ ένα μεταβατικό στάδιο δύο χρόνων ευελιξία, ώστε να μπορέσει και ο δημόσιο τομέα να ανταποκριθεί σε όλε τι απαιτήσει τη οδηγία. Εν κατακλείδη να πω ότι αυτή, ο συμβιβασμό, αυτή η νέα αναθεώρηση τη οδηγία είναι πολύ σημαντική και για την κοινωνία και για την οικονομία, ιδιαίτερα στην εποχή τη ψηφιακή οικονομία. Και θέλω να ευχαριστήσω επίση και τον πρόεδρο τη Επιτροπή, ο οποίο ε, μα στήριξε και καθ' όλη τη διάρκεια των τριών έπαιξε σημαντικό ρόλο για να επιτευχθεί αυτό ο συμβιβασμό. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους συναδέλφους. Thank you very Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσθέσουμε ότι ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις χθες τις 5 το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νεοκλή που παρουσιάσατε όλα τα αποτελέσματα, έξοχα αποτελέσματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενο σημείο συνάδελφο Ντανίκα, ορίζον Ευρώπη. Πού βρισκόμαστε πάνω σε αυτό. Πουθενά είναι η απάντηση. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν το θέμα που συζητήσαμε με το Ρουμάνο Υπουργό Έρευνας. Δεν έχουμε πρόβλημα με την Προεδρία αλλά με κάποια κράτη-μέλη. και με τις υπηρεσίες του Συμβουλίου αποφάσισαν να αμφισβητούν την νομική βάση για τις αποφάσεις. Θέλουν το Ευρωκοινοβούλιο να μην συμμετέχει στην απόφαση, να εκφράζει μόνο σύμφωνη γνώμη, να ε, εκφράζει την άποψή του και μόνο. Αυτό είναι απαράδεκτο για μας. Το μήνυμα που διαβιβάζω και διαβίβασε τον Υπουργό Έρευνας να διαβιβάσει το μήνυμα στο Συμβούλιο ε, ήταν ότι έχουμε παράλογα εμπόδια μπροστά μας. Δεν έχουμε για ποιο λόγο καθυστερεί την απάντηση το Συμβούλιο και δεν καταρτίζει κάποιο πρόγραμμα. Γιατί δεν δείχνει κάποια προθυμία να διεκπαιρεωθούν αυτοί οι δύο φάκελοι, όπως προτάθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. δεν ήταν ιδιαίτερο αίτημα. Θέλαμε να ακολουθηθούν οι συνηθισμένες διαδικασίες στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Θα σας γνωστοποιήσω περί νεωτέρων. Θα γίνει ο δεύτερος τριμερής διάλογος την επόμενη τρίτη το βράδυ. Ξεκινάμε στις 9 και στις 6 το πρωί έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος. Πολύ ωραία προβλέπονται τέσσερις τριμερείς διάλογοι και αν χρειαστεί πέντε. Στόχος εξέβρεση συμφωνίας με το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο πλευρό μας λίγο πολύ. Και όσον αφορά τη διαφορά της νομικής βάσης για την απόφαση, όταν εισηγητής είναι ο κ. Έρετ, αν πιστεύουν ότι έναντι του επομένου κοινοβουλίου θα είναι σε καλύτερη θέση, αν θέλουν να περιμένουν, κάνουν σφάλμα. Ίσως το καινούριο κοινοβούλιο, θέλει να ξεκινήσει από το μηδέν. Μπορεί να κάνουν τι θέλουν. Δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα η αναβολή για πάνω από ένα χρόνο, διότι η επόμενη Προεδρία θα μπορεί να κάνει τίποτα με αυτό το φάκελο. Δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. δεν θα υπάρχουν αυτοί που θα συμμετάσχουν στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Θα έχουμε νέο επίτροπο, λέει και ο πρόεδρο. Νέο επίτροπο και νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αλλάξουν όχι μόνο τους επιτρόπους, θα αλλάξουν το προσωπικό. Από την εμπειρία μας το 2014 είδαμε ότι είναι παράλογο να πιστεύουν την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέους επιτρόπους και τα νέα μέλη του προσωπικού. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να εργαστεί πιο πριν από τον Νοέμβριο, στην καλύτερη περίπτωση. Παράλογες καθυστερήσεις, παράλογη στάση του Συμβουλίου, επί ενός φακέλου που δεν είναι πολιτικής φύσεως, είναι τεχνικής Δεν υπάρχουν ξεχωριστές απόψεις στο Κοινοβούλιο, υπάρχει ομοφωνία. Οι λύσεις την χάνουν ευρύτατης υποστήριξης. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ποια συμβουλή σας, λέει ο Πρόεδρος, τι να κάνουμε. Να περιμένουμε μια απάντηση. Να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση. Την Τρίτη, στον τριμερή διάλογο, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή, οποιαδήποτε αλλαγή, στη στάση του Συμβουλίου και θα σας ενημερώσω τι θα γίνει. Έχουμε, έχουμε ενδεχόμενο Β και Γ στην προσέγγιση μας. Μετά λοιπόν, αφού ξέρουμε, θα σας ενημερώσουμε. Εάν υπάρξει περιθώριο επικοδομητικού διαλόγου. Αν το Συμβούλιο θα μετακινηθεί όχι, αν μπορεί να γίνει διάλογος ή όχι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Συνάδελφε μας Σαλίνη, έχουμε καλύτερες ειδήσει από την πλευρά σας. Η διαπραγμάτευσή μου είναι καλή. Είμαι ικανοποιημένος. Πρέπει να πω ότι για το διάστημα ακολουθούμε καλό δρόμο. Στο ίδιο γήπεδο έχουμε το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μικρονομικά προβλήματα για την εντολή, το καθήκον του, της νέας υπηρεσίας και τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είμαι αισιόδοξο. Μπορούμε να πετύχουμε καλή συμφωνία, κυρίω μετά τον τριμερή διάλογο. Είμαι πραγματικά αισιόδοξο. Έχουμε τεράστιο αριθμό τεχνικών συναντήσεων πριν το δεύτερο τριμερή διάλογο. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος πιθανότατα γίνεται 20 Φεβρουαρίου όπως είπα και στην προηγούμενη συνάντηση, έχουμε ισχυρή εντολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά περιμένουμε καλή εντολή και για το Συμβούλιο. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να περιμένουμε όμως. Στόχος μας, οι στόχοι μας είναι σαφέστατοι. Πρόσβαση στο διάστημα, διακυβέρνηση κλπ. συνεχίζουν οι τεχνικές συνεδριάσεις και πρέπει να πω ότι εγώ είμαι αισιόδοξο. Και όλα πηγαίνουν καλά κατά την απόψή μου. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Πριν τις εκλογές νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε για την πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ποιος είναι ο πλήρης τίτλος του προγράμματος. Η δημιουργία του διαστημικού προγράμματος της Ενώσεως και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, της Ενώσεως για το Διαστημικό Πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Υπάρχουν ερωτήσεις. Όχι. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου. Τον λόγο έχει ο κύριος Κρασνοντεύσκη, ο εισηγητής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ε, στις 16 Ιανουαρίου έγινε ήδη ο πρώτος γύρος ε, διαλόγου, σύντομος, ε, τρεις ώριτσες. Ήταν ο Ρουμάνος Υπουργός Οικονομίας, η Επίτροπος, η κυρία Μπιενκόφσκα. Ξεκινήσαμε με τα απλά άρθρα. Και βεβαίως, αν δούμε τα αποτελέσματα Βλέπω πως ε, πετύχαμε αρκετούς ε, συμβιβασμούς, ε, δηλαδή ξεκαθαρίσαμε τους στόχους, το Συμβούλιο δέχτηκε τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου σε πολλές περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποιες διαφορές απόψεων όσον αφορά κάποιες πτυχές του θέματος. Το Συμβούλιο θέλει περισσότερες περιφερειακές προτεραιότητες, το Κοινοβούλιο θέλει στρατηγική αυτονομία της Ένωσης ε, που πρέπει να τονιστεί. Αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί του θέματος. Ένα άλλο ζήτημα, ο προπολογισμό. Εδώ συμφωνήσαμε στο ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή τον προπολογισμό. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλει μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των ταμείων γιατί έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτό το ταμείο. Οπότε δεν πρέπει να μπερδεύουμε πολιτικές με στρατιωτικές δαπάνες και κάτι άλλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να έχει και έναν ξεκάθαρο προϋπολογισμό όσον αφορά τις τεχνολογίες εχμής. Και εξακολουθούν ε, εδώ οι διαπραγματεύσεις. Μετά, άλλο θέμα, εφαρμογή και οι σχετικές ε, απόψεις με τη χρηματοδότηση. Το Συμβούλιο προτείνει μια έμεση διοίκηση, μια έμεση λύση. Σύμφωνα με την αρχή του ότι σε κάποιες ε, περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το επιτρέπει. Μετά υπήρχε το ζήτημα του έμεσου κόστους και εδώ πέρα συμφώνησαν όλοι ότι ε, πρέπει να βρεθεί μια ευέλικτη λύση ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. και δεν υπάρχει κάποια συμφωνία στο τι μορφή θα πρέπει να έχει το έμεσο κόστος. Το Συμβούλιο ήθελε 50%, το Κοινοβούλιο ήθελε να έχει δύο δυνατότητες ε, υπολογισμού. να υψηλότερο όριο ή χωρίς όριο και μετά υπήρχε το ζήτημα της επιλογής των έργων. Υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά τα επιπρόσθετα κριτήρια. Το Συμβούλιο υπέβαλε μία πρόταση για τα επιπρόσθετα κριτήρια. Είναι το θέμα του επίπεδου της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Είχαμε το πρόβλημα του τι σημαίνει αυτό και αναμένουμε τώρα την πρόταση του Συμβουλίου. Τώρα γίνονται έντονες διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Στις 5 Φεβρουαρίου θα έχουμε άλλη μια συνάντηση. Και κάτι άλλο πρέπει να αναφέρω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρχε στο ίδιο το κοινοβούλιο. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν επιφυλάξεις και όχι μόνο για αυτόν τον τριμερή διάλογο. Ε, σε ποιο βαθμό μπορούμε να διαπραγματευόμαστε όταν έχουμε αποφασίσει κάποια πράγματα γενικότερα ή δεν τα έχουμε αποφασίσει, παραδείγματος χάρη, όπως το ΔΕΛΤΑΠΗ ή τρίτες χώρες, ε, το άρθρο 5. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν προβλήματα με τις αποφάσεις που έχουμε ήδη λάβει αλλά θέλουμε να ολοκληρώσουμε σε αυτήν την θητεία. Οπότε δεν έχει τώρα νόημα να το κουράζουμε. Ε, δεν θα μπορέσουμε να πούμε τίποτα συγκεκριμένα για τον προπολογισμό, αλλά θα ολοκληρώσουμε την έκθεση και τις εργασίες μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενοχλεί κάπως γιατί κάνουμε παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις. Αλλά νομίζω αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Μπορούμε να το βρούμε αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις, ε, όπως για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, έχουμε συμφωνήσει για το τι μορφή θα πρέπει να έχει η λύση ήδη από την αρχή. Είναι σαφές ότι είναι αναγκαίο και λογικό και πιθανό. Και μας λέει και η νομική υπηρεσία ότι είναι δυνατόν. Οπότε επιβεβαιώθηκε ότι θα ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό εντός του χρονικού πλαισίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ε, παρατηρήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Επιτροπή μας, για τις προοπτικές να ολοκληρωθεί κάποτε ο διάλογος. Στα μέσα Απριλίου νομίζω θα έχουμε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο θέμα, το 17, το μέσο συνδέοντα ε, την Ευρώπη. Τον λόγο κυρία Βίρκουνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινήσαμε χθε του τρίμπερι διαλόγου. Ήταν η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Όπω ξέρετε, έχουμε κοινή έκθεση μεταξύ Επιτροπών Ρήτρα και Τραν. Δεν αναμένω ότι θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα γιατί πιστεύω ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι αρκετά κοντά στι θέσει τους χθες επικεντρωθήκαμε κυρίως ε, στα θέματα μεταφορών και σε κάποια οριζόντια θέματα και την επόμενη εβδομάδα στις τεχνικές ε, συνεδριάσεις θα συζητήσουμε τα θέματα τα ενεργειακά και τα ψηφιακά, αλλά δεν περιμένω στα ψηφιακά να έχουμε μεγάλες δυσκολίες ε, στην ενέργεια. Έχουμε τα νέα διασυνοριακά προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και είχε προτεθεί ότι το 10% του Ταμείου για την Ενέργεια να χρησιμοποιείται για τις ανανεώσιμες ε, στην ε, Ολομέλεια φτάσαμε στο 20% για τα διασυνοριακά αυτά τα προγράμματα και επίσης ε, έχουμε και κάτι μεγαλύτερο από αυτό το της Κομισιόν, μιλάμε για 15%. Θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν. Τώρα, Σκοπεύουμε να έχουμε δύο ακόμη τριμερείς διαλόγους και θα έχουμε μία μεικτή συνεδρίαση των Επιτροπών Τραν και Ήτρε το Μάρτιο και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τότε αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Απριλίου. Είχαμε όμω τώρα μόνο έναν τριμερή διάλογο, αλλά σχεδιάζουμε πολλέ τεχνικέ συναντήσει. Τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμβασμού. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Αυτά. Ωραία. Να ό,τι κατάλαβα η πρώτη χτεσινή συνάντηση του τριλόγου αφορούσε κυρίως ε, τις μεταφορές ε, και οι επόμενες συναντήσεις θα αφορούν θέματα της Επιτροπής Ήτρε. Ο κύριος Μαρινέσκου μάλιστα είναι υπεύθυνο ε, της Επιτροπής Μεταφορών, καθώς ε, είναι και πλήρες μέλλον της Επιτροπής. Ήταν πολύ καλό αυτό για μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν Χένα για την παρουσίασή σας και ελπίζω όλα να πάνε ομαλά και γρήγορα για να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα σε αυτή τη θητεία. Επομένως, ολοκληρώσαμε και το 17. Πάμε στο 18 τη σημερινή διάταξη ανταλλαγή απόψεων με τον Τζουλιάν Κίνγκ Ευρωπαϊκό Επίτροπο Αρμόδιο για την Ένωση ασφάλεια σχετικά με τον προπολογισμό για την έρευνα στον τομέα τη ασφάλεια στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μα, κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε τον προπολογισμό για την έρευνα στον τομέα τη ασφάλεια, ε, υπό το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους πολίτες. Θα θέλαμε να μας πείτε κάτι σχετικά με τα αποτελέσματα και την κατάσταση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας και το ESRP χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και το πρόγραμμα Horizon 2020. 7ο πρόγραμμα πλαίσιο λοιπόν, Horizon 2020 είναι το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο όπως ξέρετε. Και έχετε, έρχεστε σε μια πολύ καλή χρονική στιγμή, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον οριζόντα Ευρώπη. Και βέβαια συζητάμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο που είναι κάτι διαφορετικό, αλλά όχι και τόσο διαφορετικό όταν συζητάμε το Ταμείο Άμυνας για την βιομηχανία μας ή όταν συζητάμε τον προϋπολογισμό για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας στο πρόγραμμα πλαίσιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Πίτροπε. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για την ευκαιρία να συζητήσω με αυτή την Επιτροπή. Γνωρίζω ότι μιλάω σε μέλη με βαθιά τεχνογνωσία επ' αυτών των θεμάτων και ελπίζω να μάθω κι εγώ κάτι από αυτή την συνομιλία, όπως και οποιοδήποτε άλλος. Ευπρόσδεκτη ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα μαζί σας. Είναι θέμα ενδιαφέρον σας απασχολεί. Σημαντική αυτή η ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω, ελπίζω λέγω, ότι θα ανακαλύψουμε ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Με αυτή την ελπίδα λοιπόν, ας δώσω το εναρκτήριο λάκτισμα και να κάνω ένα βήμα πίσω και να κοιτάξω μπροστά. Ξέρω τι ξέρετε, διότι έχω μιλήσει με κάποιους από εσά, αντιμετωπίζουμε περίπλοκο, μετακινούμενο, μεταλλασσόμενο πρόβλημα απειλής. Ένα περιβάλλον μεταλλασσόμενο απειλής. Επεξεργάζουμε το θέμα δυόμιση χρόνια και όλες οι πτυχές του έργου που κάνουμε για την Ένωση Ασφάλειας, καταπολέμηση τρομοκρατίας, αντιμετώπιση ριζοσπαστικοποίησης, κλασική κυβερνοασφάλεια, κυβερνοαπειλές που στρέφονται κατά των συστημάτων μας, κατά των πλατφορμών μας, κατά των υποδομών μας, είτε είναι αυτά, είτε είναι καινούριες απειλές που έρχονται από τον κυβερνοχώρο, κακή χρήση, αρνητική επιβλαβής χρήση των διασυνδέσεων μας με το διαδίκτυο, να μας βλάψουν, να απειλήσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και τους δημοκρατικούς θεσμούς και μη λησμονούμε και το οργανωμένο έγκλημα. Όλα αυτά είναι μέτωπα. Και σε αυτά τα μέτωπα αλλάζει συνεχώς η εικόνα της απειλής, εξελίσσεται και πρέπει και εμείς δεόντως να αλλάζουμε τις απαντήσεις μας. Όσο με αφορά, η έρευνα για τα θέματα ασφαλείας είναι ένα απόσπαστο τμήμα της προσπάθειας. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε κατάλληλους πόρους, να διοργανώσουμε σωστά τον τομέα, να δούμε στο μέλλον πώς πρέπει να διεξάγεται αυτή η μελέτη. Ευχαριστούμε την Επιτροπή σας και την προσπάθεια που καταβάλλετε, τον ενδιαφέρον που δείχνετε, που θεωρώ ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, πώς θα δημιουργήσουμε έρευνα για την ασφάλεια που προστατεύει τα συμφέροντά μας έναντι των μεταλλασσομένων απειλών. Πρέπει να είμαστε πάντα επίκαιροι έναντι των απειλών και των προκλήσεων που συνεχώς αλλάζουν, άρα χρειαζόμαστε έρευνα για θέματα ασφαλείας που έχει συγκεκριμένους σωστούς στόχους, καλύπτει τις ανάγκες εκείνων που προσπαθούν να επιβάλλουν την ασφάλεια των δυνάμεων επιβολής του νόμου και εκείνων που διαμορφώνουν την πολιτική. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ελπίζω να συμφωνείτε λόγω του βάρους και της σημασίας που έχουν τα χρήματα που διατίθεται για την έρευνα. Δύο δισεκατομμύρια την περίοδο που αναφέρατε, αυτό είναι περίπου το ίμιση όλης της δημόσιας χρηματοδοτήσεως για την ασφάλεια, την έρευνα για την ασφάλεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ψηλότερο ποσοστό από ό,τι σε άλλου ερευνητικού τομεί. Το πρόγραμμα ορίζουν συνολικά είναι 10 με 15% έναντι 50%. Άρα, στην πράξη υπάρχουν κράτη-μέλη που εξαρτώνται σχεδόν απόλυτα από την έρευνα, τη χρηματοδότηση για την έρευνα περί ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να πραγματοποιήσουν τη δική τους έρευνα ασφαλείας. Άρα έχουμε ε, υποχρέωση να είμαστε σωστοί, να οργανώσουμε σωστά αυτή τη χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Horizon. Χρειάζεται λοιπόν να οργανωθεί έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, θα πρέπει να, τα αποτελέσματα να αυξηθούν, να αντιμετωπίσουμε έτσι διασυνοριακά και υπερεθνικά προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια και αν γίνει σωστή δουλειά να εξασφαλίζουμε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών θα είναι διαθέσιμα ε, σε όλη την Ένωση. Η προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσης επιτρέπει να τηρήσουμε και να αναπτύξουμε επιτυχή βιομηχανία αμυντική και ασφαλεία στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια προβλήματα να διαφυλαχθούν θέσει απασχόληση και να συμβάλλουμε και στην αυτόνομη δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω όσον αφορά τον τομέα τη ασφάλεια. Για αυτού του λόγου, οι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Προγράμματα όσον αφορά ε, μέθοδος για συλλογή ηλεκτρονικών στοιχείων, ε, ιατροδικαστικά στοιχεία κλπ. Είναι ζωτική σημασία αυτή η δουλειά όχι μόνο να συνεχιστεί και στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο, αλλά στο βαθμό του δυνατού να ενισχυθεί βάσει των προτάσεων για τον ορίζοντα Ευρώπη. Και αυτό ελπίζω να σας βρίσκει συμφώνους. Τα ερευνητικά μας προγράμματα την ασφάλεια εστιάζονται σε τρεις τομείς. Κοινωνίε που αντέχουν στι καταστροφέ, αντιμετώπιση χημιολογικών, βιολογικών, ραδιολογικών, πυρηνικών απειλών, προστασία και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένη και στην αντιμετώπιση τρομοκρατία και κυβερνοασφάλεια. Στον τομέα Τη αντοχή έναντι καταστροφών πρέπει να συνεχίσουμε τη βελτίωση της δυνατότητα να εμποδίσουμε, να ανταποκριθούμε και να ανοικοδομούμε μετά από καταστροφές, φυσικές καταστροφές φερρυπίν, πυρκαγιές καταστροφικέ, όπω είδαμε σε πολλά κράτη-μέλη πρόσφατα το, καλοκαίρι, όπως ε, επιθέσεις χημικές που κατά παρελθόν θεωρούσαμε ότι δεν πρόκειται να συμβούν, αλλά ξέρουμε ότι στο Σόλσμπερι τι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι είναι δυνατές αυτές οι επιθέσεις, θα πρέπει να βελτιώσουμε την προστασία και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων και των κρίσιμων υποδομών. Υπάρχει ζήτηση πραγματική από τις αρχές, όλα τα κράτη-μέλη και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τις δημοτικές αρχές να συνεργαστούμε μαζί τους για καλύτερη ε, αντοχή που θα, και προστασία των δημοσίων χώρων. Χρειαζόμαστε καινοτόμε λύσεις γιατί έχουν προβλήματα που αυξάνονται στον κυβερνοχώρο, δεν χρειάζεται να σα το πω, έγινε αλλαγή ρυθμού όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, όσον αφορά τους, τις και υπάρχει ζήτηση από τα κράτη-μέλη συνεργασίας μαζί μας για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες επιθέσεις στο διαδίκτυο. Εκεί θα πρέπει να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες Επίσης πρέπει να βελτιώσουμε και την κατανόηση και την αντίληψη των ανθρωπίνων παραγόντων. Τι κρύβεται πίσω, ποια κίνητρα υπάρχουν, τι οδηγεί ένα νέο να γίνει ριζοσφαστικοποιημένος. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι αποτελέσματα έχουν τρομοκρατικές επιθέσεις, πώς να ανταποκριθούμε, να δίνουμε πρώτη απάντηση στις επιθέσεις και να φροντίζουμε και τα θύματα. Πρέπει να ακούμε και τους πολίτες και να μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν στην έρευνα που κάνουμε την ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε ότι οι καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύσσονται με έναν τρόπο είναι συμβατός με τις προσδοκίες τους και να τους διαβεβαιώνουμε ότι πάντα αυτό θα γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ιδιωτικότητα και δοντολογικά πλαίσια. Διότι επιτυχής πολιτική ασφαλείας θα πρέπει να εδράζεται επί του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλιώ αρχίζει να χάνει κανείς τη στήριξη του λαού. Μπορούμε να βελτιώσουμε τις, τα αποτελέσματα τη έρευνα για την ασφάλεια, να ενταχθεί σε μια διαδικασία δημιουργία δημιουργικότητα, εντοπίζοντα τι ανάγκε για να εφαρμόζονται οι λύσει. Θα πρέπει διαμορφώνοντα την πολιτική, οι δυνάμει του νόμου, οι δυνάμει πρώτη αρρωγή, οι τη πολιτική να αναπτύσσουν τι αναγκαίε δυνατότητε, αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών. Υπό το παρόν πρόγραμμα Horizon 2020, τα προγράμματα ερευνητικά πρέπει να συμπεριλαμβάνουν του ειδικού, αυτού που εφαρμόζουν τα μέτρα. Αυτό υπήρξε επιτυχέ, βοήθησε να ευθυγραμμίσουμε την έρευνα με τι ανάγκε εκείνων που εφαρμόζουν τα μέτρα επιτόπου και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Επίση, φρονώ ότι οι διάφορε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, που είναι επιτυχέστατε στον τομέα, η Europol, Φερρυπίν, η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και η Μεθοριοφυλακή θα πρέπει να συμμετέχουν εντοπίζοντα τι ανάγκε που πρέπει να αναπτύξουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να δίνουν συμβουλέ όσον αφορά την ανάπτυξη των προγραμμάτων, τι ανάγκε των χρηστών και να παίζουν και ένα ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων τη ε, έρευνα. Βλέποντα ποια είναι η παρούσα κατάσταση όσον αφορά τον ορίζοντα 2020, συνεχίζονται οι συνομιλίε διοργανικέ. Η Επιτροπή ε, πρότεινε να έχουμε και διαφορετικές συναθρήσεις μονάδων κοινωνικών και προτείνεται να προσθέσουμε λεπτομέρειες όσον αφορά τις δραστηριότητες που καλύπτονται τομείς παρέμβασης για την προστασία των συνόρων, διαχείριση των συνόρων, πειρατεία, ε, παραποιημένα προϊόντα, υποστήριξη της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης για την πρόληψη συγκρούσεων και την ε, ε, ε, ειρήνευση. Όπως σας είπα, από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουμε ξεχωριστή συστάδα μέτρων που καλύπτονται αυτές ε, οι μονάδες οι κοινωνικές που δημιουργούν την ασφάλεια και τις σχετικές δραστηριότητε τις υποστηρίζουμε με πάρα πολύ ανοιχτό πνεύμα. Όσον αφορά τις περαιτέρω προτάσεις Επιτροπής, αυτό το θέμα για τις ασφαλείς κοινωνίες, αυτό το τμήμα θα πρέπει να υπάρχει το 2% από τον ορίζοντα από ό,τι κατάλαβα θα πρέπει να περιμένουμε για τα αποτελέσματα όμως των διοργανικών συζητήσεων για το γενικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε πρόταση και έκθεση του Κοινοβουλίου είναι έξοχη βάση για σωστή επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα περί ασφαλείας στο μέλλον. Τέλος, επειδή τα αναφέρατε και ξέρω ότι είναι ένα θέμα που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην Επιτροπή σας, να αναφερθώ στο θέμα της αμυντικής έρευνας. Το ορίζον Ευρώπη όπως ξέρετε άριστα παρέχει νομική βάση για την αμυντική έρευνα και τα σχετικά προγράμματα, διότι προβλέπεται αυτό από τη συνθήκη, όμως παρόλα αυτά θα αποτελέσει τμήμα ξεχωριστού ταμείου για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, και θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες για αυτό το ταμείο και θα πρέπει η χρηματοδότηση να είναι περίπου πάνω, θα είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια ε, ευρώ χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Υπάρχουν συνεργασίες που δημιουργούνται μεταξύ Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου από τη μια πλευρά και του Ορίζον Ευρώπη από την άλλη. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι και οι δύο τομείς, πολιτικός και στρατιωτικός, θα ωφεληθεί, δεν θα υπάρχει επικάλυψη όσον αφορά την έρευνα, αλλά βασικά συμφωνούμε με αυτό που θεωρώ ότι είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Να κλείσω λέγοντας ένα ευχαριστώ προς το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα σε αυτή την Επιτροπή για τη δουλειά που κάνετε, για την συνεχές ενδιαφέρον και υποστήριξή σας, για την έρευνα περί ασφαλείας του προγράμματος που κάνει πραγματικά τη η διαφορά βοηθά να έχουμε κάπως πιο ασφαλείς και σίγουρους τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την σαφή σας τοποθέτηση και ανοιχτή επίσης. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται για την χρηματοδότηση της ασφάλειας και την έρευνα στον τομέα της άμυνας. Αν μου επιτρέπετε, ερωτήσεις από το ΕΛΚ. Ναι, ο κύριος Έιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε για τα όσα είπατε, αλλά κυρίως για τα όσα κάνετε τα τελευταία χρόνια που δείχνουν το τι απώλεια είναι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα δούμε τι θα γίνει. πάντων, στην ουσία. Εκτιμούμε έτσι αυτό, την πόκα που παίζουμε με τα φιλικά ψέματα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Είναι η τρίτη φορά που φτιάχνουμε ένα συγκεκριμένο τέτοιο πρόγραμμα έρευνας. Και είναι απολύτω λογικό ο διαχωρισμός από το υπόλοιπο πλέγμα. Θα ήθελα τώρα να προσθέσω και εγώ κάτι στο θέμα. Ήδη αναφέρατε ότι υπάρχει ένας ε, τομέας παρέμβασης ε, στο, στην προστασία των συνόρων υπό το φως των αποφάσεων Συμβουλίου και Κομισιών. Αναφέρατε επίσης την πειρατεία και την κυβδηλία προϊόντων για προφανείς λόγους. Πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη απώλεια για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεύτερον, είναι μια απειλή την οποία δεν έχουμε αντιληφθεί πλήρως καθώς οι ειδικοί υπολογίζουν ότι ένα 4% των ευρωπαϊκών φαρμάκων που πολλούνται είναι ε, κάποια ε, περίεργης ε, κατασκευή και προελεύσεως. Και η τρίτη πτυχή είναι ότι βλέπουμε γιατί το θεωρούμε ως ένα έγκλημα χαμηλού κινδύνου αλλά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς αποδίδουμε έμφαση σε αυτό. Αυτό το οποίο δεν αναφέρατε αλλά έχει κάποια σημασία είναι ακριβώς η προώθηση του συντονισμού, της συνεργασίας και ανανεώσαμε την πρότασή μας και είπαμε ότι θα έχει νόημα να συνεργαστούν περισσότερο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τώρα θα είναι όργανα της Κομισιόν και ευρωπαϊκά όργανα όπως η Europol γιατί θεωρούμε ότι δεδομένου του ότι έχουμε ένα πρόγραμμα έρευνας κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων και χρηματοδοτούμε το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Europol με κάποια σχετικά πενιχρά ποσά, 5 με 10 εκατομμύρια ευρώ, αναλόγως με το πόσο τα μετράει κανείς. Έχει νόημα ε, να συγχωνευτούν αυτά τα θεσμικά όργανα και να σκεφτούμε να πάει ένα μέρος αυτών χρημάτων σε αυτό το θεσμικό όργανο το οποίο θα μπορούσε να βοηθηθεί από την ε, έρευνα και ανάπτυξη από την δική σας γενική διεύθυνση αλλά πρακτικά νομίζω ότι θα ήταν λογικό να δώσουμε και προπολογισμού σε θεσμικά όργανα όπως η Europol κάτι το οποίο δεν γινόταν όχι για λόγους των Υπουργείων Εσωτερικών, αλλά για λόγους των Υπουργείων που είναι αρμόδια για την έρευνα, γιατί θεωρούσαν ότι χάνουν μια αρμοδιότητα. Έτσι λοιπόν η Europol πραγματικά χάνει την ευκαιρία να κάνει έρευνα κοντά στην αγορά, που βεβαίως ε, εδώ πέρα δεν μιλάμε για αγορά, γιατί μιλάμε για δημόσιους φορείς αποκλειστικά, οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε. Και ε, τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στον προϋπολογισμό. Αναφερθήκατε στο 2%. Το 2% σημαίνει αύξηση του προϋπολογισμού ούτως ή άλλως, ουσιαστική. Οπότε είχαμε ένα ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ ανά περίοδο και τώρα θα υπάρξει μια αύξηση αρκετά σοβαρή και αντιλαμβάνομαι ότι η Κομισιόν και Συμβούλιο έχουν την θέση ότι πρέπει να δοθεί βάρος στο πρόγραμμα έρευνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο καθηγητής Κασνοντεύσκη. Έχω μια ερώτηση για το θέμα που θέσατε στην παρουσίασή σας και συγκεκριμένα τη διάκριση που είναι σημαντική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ της έρευνας για σκοπούς άμυνας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και του Ορίζον Ευρώπη. έχω μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό να έχουμε αυτή τη διάκριση. Γιατί όταν εξετάζουμε ότι το κλασικό προϊόν της αμυντικής βιομηχανίας, τα αν ξεροπλάνα κτλ. Άρα τώρα μιλάμε για το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνό χώρο. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Γιατί υποθέτω ότι πολύ από την έρευνα που θα γίνει για το Horizon Ευρώπη θα είναι σχετική να χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς άμυνας. Πιστεύετε ότι στην πράξη, στο μέλλον, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Μπορούμε να τη διατηρήσουμε. Νομίζω ότι για το Κοινοβούλιο ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε σαφή διάκριση μεταξύ του κοινωνικού ταμείου, του ταμείου συνοχής, να μην έχουμε δηλαδή χρήματα που να μην χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας, όμως για το ρίζον Ευρώπη, σε αυτούς τους νέους τομείς όπως η ασφαλεία στον κυβερνοχώρο. χώρο. αναφέρεται και αυτή την ε, τάση δημοκρατικής επιρροής στα κράτη-μέλη. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθεί μια τέτοια κανονική διάκριση, αλλά θα ήθελα την προσωπική σας άποψη από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούμπιχ. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Αυξάνονται οι απειλές και μάλιστα με δυναμικό τρόπο. Εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε την Επιτροπή ΣΤΟΑ. Έχουμε την αξιολόγηση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών στη ΣΤΟΑ. Έχουμε κάνει κάποιες μελέτες για το πώς χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι, οι ψευδείς ειδήσει, η πληροφόρηση και ίσως είναι ζωτικό αυτό το θέμα. Γιατί αυτές οι δραστηριότητες πολύ γρήγορα γίνονται viral και φυσικά με τις ψευδείς ειδήσει βλέπουμε ότι σοβαροί πολιτικοί μπαίνουν σε σοβαρά προβλήματα. Τώρα, αν τρέξουμε το Ρίζον Ευρώπη, Ε, όταν μιλάμε για δραστηριότητε ασφάλεια, ε, τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα και την κυριότητά του. Ξέρετε ότι δεν έχουμε κυριότητα όταν μιλάμε για τη χρήση των κινητών μα. Γιατί μπορεί να έχουμε 60 σελίδε γενικών κανόνων ε, και αν ανοίξει. Παραδείγματο χάρη μια εφαρμογή, μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο, την κάμερα, μπορεί να κάνει τα πάντα στο τηλεφωνό σου χωρίς ε, να πάρεις καμία πληροφορία. Έχουμε το MIT στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα νέο πανεπιστημιακό τμήμα που προσπαθεί να κατανοήσει ποιο κατεβάζει και ποιο ανεβάζει τα δικά μου δεδομένα και τα δικά σας δεδομένα. Και δεν ξέρουμε καθόλου τι δεδομένα συλλέγουν. Και πώς στη συνέχεια πολλούνται τα δεδομένα αυτά. Αν παραδείγματο το ε, χάρη, ε, λείψουν, ε, εξαφανιστούν ε, κάποιες ε, διευθύνσεις στο ηλεκτρονικό δρομείο, μπορεί κάποιος να τις έχει υποκλέψει. Για την προστασία των δεδομένων, θα ήθελα να ξέρω ποιος αλγόριθμος χρησιμοποιείται για τα δικά μου δεδομένα. Και υπάρχει περίπτωση να έχουμε χαρτογράφηση των αλγορίθμων. Δηλαδή, οι αλγορίθμοι να μην είναι διαθέσιμοι για μία μικρή ελίτ εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δυνατόν να τα έχουμε και εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα ευρύ πρόγραμμα ανοιχτή επιστήμη, που να μπορεί να ενημερώνει του ανθρώπου τι γίνεται ε, στα παρασκήνια στη χρήση, κατά τη χρήση αυτών των συσκευών. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη και χρειαζόμαστε και διαφάνεια στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. να έχετε το λόγο. Ναι. Θέλω να προσθέσω μια ερώτηση. Θα μας βοηθούσε να ξέρουμε ποιες είναι οι ιδέες σας για το πρόγραμμα. Στο πρώτο πρόγραμμα 1,3 δις ξοδέψαμε. Στο πρόσφατο 1,7 δις. αν ακολουθήσουν πρώτα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αύξηση που προβλέπεται από το Κοινοβούλιο, πάμε στα 2 δι ευρώ περίπου για αυτό το πρόγραμμα. Δεν θέλω να βάλω φωτιά στο θέμα. Αν δίνατε 2 δισεκατομμύρια στο Europol, θα ήταν μεγαλύτερη αστυνομική οργάνωση στον κόσμο. Στα όρια των, της εντολής της. Ερώτηση μετά από δύο προγράμματα. Πώς τα αποτελέσματα των προγραμμάτων πλησιάζουν περισσότερο την πραγματικότητα. Πάντα είναι δύσκολο να αναλύσουμε παρκώς την ασφάλεια. Τι ιδέα έχετε σχηματίσει. Το Europol έχει 5-6 εκατομμύρια για ασφάλεια, για το κέντρο ασφάλειας Και το πρόγραμμα περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ για την κυβερνοασφάλεια, για την έρευνα. Επιτόπου, πώς υλοποιούνται, πώς εφαρμόζονται, ποια είναι η εμπειρία σας όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα και μελλοντικά ποιο είναι το όραμά σας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Να προσθέσω κι εγώ ένα σχόλιο ή ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ασφάλεια και το σχετικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες εκατομμύρια, χιλιάδε χιλιάδες προγράμματα μόνο. Στα πλαίσια του 7ου και 8ου προγράμματος πλαίσιο. Το πιο δημοφιλές αρχικά ήταν οι τεχνολογίες διπλής χρήσεως. Ασφάλεια και να βοηθήσουμε και ανθρώπους με κάποια αναπηρία και το ονομάσαμε πρόγραμμα διπλής χρήσεως. Αν θέλουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ άμυνας και ασφάλειας, ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε τις τεχνολογίες διπλής χρήσεως αυτή τη φορά. Εδώ ασφάλεια και άμυνα είναι η διπλή χρήση. Θα ήταν ένας νέος τύπος διπλής χρήσεως. Όχι για χρήση στον πολιτικό τομέα, αλλά για την ασφάλεια. Λοιπόν, αυτό θα ήταν μια καλή λύση. δεν θα αναπτύσσετε μια, μια λύση για ασφάλεια και άμυνα ξεχωριστά. Είναι πιο καλό να έχουμε μια τεχνολογία και να εφαρμόζουμε σε δύο τομεί αντί να αναπτύσσουμε δύο ξεχωριστέ τεχνολογίε. Διπλή χρήση. Νέο τρόπο, νέα φόρμουλα για διπλή χρήση, όπω τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Ε, έχετε το λόγο, Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα όπου επικρατεί σαφήνεια και κάποια που θα πρέπει να αποσαφινιστούν με τις συζητήσεις μας. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ο διαχωρισμός των διαφόρων αυτών ε, κόμβων, των κλάστερ, είναι καλή ιδέα. Και έτσι θα βρεθούν τα σωστά προγράμματα με το διαχωρισμό. Η διαδικασία συνεργασίας και συνεργασίας με τους εμπλεκομένους φορείς για την κατανομή των προγραμμάτων. Όπως ξέρετε, πολύ καλά, είναι η διαδικασία χρονοβόρα. Όποιες απόψε εκφράζω σήμερα είναι προσωπικές. Δεν δεσμεύεται κανείς εκτός από μένα. Διότι θα ακολουθεί την πορεία της η διαδικασία. Πιστεύω ότι οι τομείς που ανέφερα είναι τομείς που πρέπει να στοχεύουμε. Θα υπάρξουν και άλλοι τομείς, πέραν από αυτούς, που θα διαφανούν τι τις συζητήσεις. Κύριε Έλερ, από δύο σκοπιές εξετάσατε ένα τομέα. Τη στήριξη προς τις υπηρεσίες. Ανέφερα τις υπηρεσίες ξεχωριστά. Όχι μόνο τις γνωστές όπως είναι η Europol ή την ακτοφυλακή και τις μεγαλύτερες, αλλά ένα φάσμα υπηρεσιών που δημιουργήσαμε πρόσφατα στον τομέα της ασφάλειας και που δημιουργούμε, κυρίως όσον αφορά τον κυβερνοχώρο. Αυτές οι υπηρεσίες έπρεπε να παίζουν μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά την έρευνα που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Προσωπικά είμαι ανοιχτό για το πώς μπορεί να κινηθούμε. Τι θα κάνουμε, να πλησιάσουν οι υπηρεσίες τις μορφές των προγραμμάτων και την υλοποίησή τους στις παρούσες δομές ή άλλη λύση που προτείνατε. Να τους δίνουμε χρήματα. Αυτά τα ταμεία μπορούμε να το συζητήσουμε. Τι θα έλεγα. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι οι υπηρεσίες ασφαλεία στερήθηκαν χρηματοδότηση. γίνονται συζητήσεις, πολύ συχνά με τη στήριξη του Κοινοβουλίου και συζητήσεις συχνά καταλήγουν σε μια καλή ρύθμιση χρηματοδοτήσεως για τις υπηρεσίες μας. Και αυτό είναι πολύ σωστό, διότι κάνουν πολύ σημαντικό έργο. Όμω, εντάξει, ας δούμε πώς μας συμμετέχουν περισσότερο τώρα από ό,τι κατά το παρελθόν υπηρεσίες στην έρευνα και ανάπτυξη. Τώρα, σχέση μεταξύ άμυνας, ασφάλειας και πολιτικού τομέα. Η σχέση αυτή πρέπει να εξεταστεί. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το συμπέρασμα. Χρειάζεται εξέταση όμως. Και αυτό στα πλαίσια του κυβερνοχώρου. Και αυτό αφορά μια σειρά ερωτήσεων που θέσατε. Τι έχουμε λοιπόν. Τον ορίζοντα Ευρώπη, το ETF, το Αμερικό Ταμείο και το Digital Europe, το Ταμείο για την Ψηφιακή Ευρώπη. Και όσον αφορά τον κυβερνοχώρο, υπάρχουν κάποιες ατάξεις για τον κυβερνοχώρο στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Ταμείο ολοκληρωμένη Διαχείρισης Συνόρων, επιδιώκοντα την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο διεξαγωγή συζητήσεως περί σεβασμού των διαφόρων σκοπών, των διαφόρων ταμείων από τη μια και τη φύση τους και από την άλλη συντονισμένη, ολοκληρωμένη υποστηρικτική προσέγγιση προς την έρευνα και την ανάπτυξη για τον κυβερνοχώρο και μάλιστα να ελέγξουμε και που υπάρχουν επικαλύψεις. Μπορεί να υπάρχει επικάλυψη μεταξύ πολιτικού τομέα, ε, εσωτερικής ασφαλείας και άμυνας. Δεν έχω απάντηση. Είναι ένας τομέας που πρέπει μαζί να κινηθούμε και να συζητήσουμε με την πάροδο του χρόνου. Το μεταξύ του EDF και του Horizon Ευρώπη. Το EDF κατά την άποψή μου πρέπει να εστιάζεται στην αμυντική έρευνα. Και υπάρχουν κάποια στοιχεία αμυντικής έρευνας στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν και θέματα και στοιχεία διπλής χρήσης. Το ορίζον Ευρώπη, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ασχοληθεί με την υποστήριξη της τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας και βιομηχανικών δυνατοτήτων. Πρέπει να εξεταστούν οι κίνδυνοι πώς μειώνται οι κίνδυνοι όσον αφορά νέες και μελλοντικές ψηφιακές τεχνολογίες. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό, μεγάλο θέμα. Δεν αφορά πτυχές του, του κόσμου όπως είναι σήμερα διασυνδεδεμένος. Είναι τα blockchains, είναι η τεχνητή νοημοσύνη και διάφορα άλλα. Πρέπει να δώσουμε και δυνατότητα στις δημόσιες αρχές, τους πολίτες, και τον ιδιωτικό τομέα να προστατεύουν τα στοιχεία τους. Απαντώντας τον κύριο Ρούτολ αυτό, να προστατεύουν τα δεδομένα τους και τις ε, δραστηριότητες τους στο διαδίκτυο. Όλα αυτά πάντα κάνουμε στο πλαίσιο του Horizon Ευρώπη. Έχουμε και κάποια χρήματα, όπως τα είδατε, που χορηγούνται για την κυβερνοασφάλεια στην ψηφιακή, στο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, Digital Europe. Κάτι που υποστηρίζω ένθερμα. Και η Μαρία Καμπριέλ και άλλοι επίτροποι είναι, υποστηρίζουν το θέμα αυτό. Δεν είναι λειτουργικός διαχωρισμός, αλλά συριακή ακολουθία δραστηριοτήτων. Το ρίζον Ευρώπη να επί και έρευνας, και ανάπτυξη δυνατοτήτων. Η διάθεση στην αγορά, η υλοποίηση, εφαρμογή πρέπει να είναι στόχος περισσότερο του Digital Europe και της χρηματοδοτήσεως που έρχεται από εκεί. Σε κάποιες περιπτώσεις όπου κανείς εργάζεται συνεργαζόμενος με την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν αφορά την Ευρωπόλπη συγκεκριμένα, ίσως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας αν τώρα είναι με τα σύνορα και την ακτοφυλακή, ε, το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων. Πρέπει να δούμε τις διάφορες πηγές χρηματοδοτήσεως που υπάρχουν για την κυβερνοασφάλεια με έναν κοινό φακό. Τα ταμεία έχουν ειδικού σκοπούς στον τομέα μας αυτό, επειδή είναι οριζόντιος, διασχίζει τους διάφορους τομείς, καλύπτει του διάφορους τομείς, και επειδή όλα αλλάζουν κατά τη διάρκεια ζωής των προγραμμάτων, γι' αυτό χρειάζεται μία αέναη προσέγγιση, με λογική προσέγγιση, όσο μπορούμε. Εδώ δεν αποφεύγω τις ερωτήσεις, πραγματικά νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος όπου συνεργαζόμενοι θα σημειώσουμε πρόοδο για να αναπτυχθεί η κυβερνοασφάλεια, οι δυνατότητες που έχουμε κυβερνοασφάλεια, θα υπάρξει ζήτηση και απέτηση να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι βέβαιο και να αντικατοπτρίσουμε το τρόπος την μεταλλασσόμενη φύση των απειλών που θα αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί απόλυτα, κυρίως την τελευταία ομάδα ερωτήσεων. Αυτή είναι η άποψή μου όμως για το φάσμα των θεμάτων που ετέθησαν. Σας χαιρετίζω για τη συνεχή υποστήριξη που παρέχεται σε μας για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε την έρευνα σε αυτόν τον τομέα και να τη χρηματοδοτούμε σωστά, γιατί πιστεύω ότι κάνει τη διαφορά, συμβάλλει σημαντικά, είτε στους τομείς εχμής που προαναφέραμε, είτε σε πιο παραδοσιακούς τομείς, να προστατεύει κανείς τα σύνορα καλύτερα, Φερρυπίν. Δεν ξέρω αν είναι κάτι παραδοσιακό ή όχι, αλλά γίνεται απαιτούμενο, πρακτική απέτηση, πώς αντιμετωπίζει κανείς τα μη επανδρομένα επτάμενα οχήματα, τα drones και πώς αυτά παρεμβαίνουν στην ασφάλεια, πώς δημιουργούν θέματα ασφαλείας και πώς κάνεις την απαιτούμενη κοινωνική έρευνα για να αντιμετωπίσεις το θέμα της ρίζος πρακτικοποίησης είτε είναι από εξτρεμιστές στο Τσάντ που γίνεται αυτό ή βίαιους εξτρεμιστές της άκρας δεξιάς, της άκρας αριστεράς. Υπάρχει ένα φάσμα προσπαθειών που πρέπει να γίνουν που είναι σημαντικότατες ούτω ώστε να πετύχουμε μια ένωση ασφαλείας, κάτι που μας ζητούν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ήταν πολύ σημαντικό να συζητήσουμε όλες τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των ε, διάφορων μερών. Είναι πολύ σημαντικό που μας ε, τα εξηγήσατε όλα αυτά. Θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ κύριε Έλερ. Εφόσον έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ιστορικό. Ορθά είπατε. Και μπορούμε να το σκεφτούμε αυτά, αλλά ο λόγος Όταν ε, λέμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τα πρωτότυπα και να διευκολύνουμε το τεστ και ε, λύσεις ε, πρώτης αγοράς, ε, αυτό προέρχεται από το δίκαιο ανταγωνισμού. Είναι πολύ πιο εύκολο υπό τον ΠΟΕ να έχουμε προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρχει ένα πρόγραμμα έρευνας. Και Υπάρχει κάποιος λόγος λοιπόν που σχετίζεται με το δίκαιο ανταγωνιστικότητας και συναφή ζητήματα. Για ποιο λόγο είναι πιο εύκολο αυτό να το εκτελέσουμε με χρηματοδότηση για την έρευνα μέσω ενό ειδικού προγράμματο έρευνα παρά με άλλο τρόπο. Επί τη ουσία, δηλαδή είναι κάτι που μπορούμε να το σκεφτούμε, αλλά δεν θέλαμε να στραφούμε σε άλλου τομεί. Υπήρχε ένα πολύ τεχνικό λόγο που το κάναμε αυτό. Και Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να σας επισημάνω, γιατί θέλω να είμαι σίγουρη ότι εσείς και η Γενική σας Διεύθυνση παρακολουθείτε τις διαπραγματεύσεις, όπου η Κομισιόν θα παίξει σημαντικό ρόλο ως διαιτητής μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Το προωθούσαμε αυτό είχαμε ορίσει την πρόθεση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ακροτήτων ε, σε ε, διάφορες μη στρατιωτικές αποστολές και τεχνολογική ανάπτυξη για να χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες για να αυξήσουμε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν να βρούμε συμφωνία εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά δεδομένης της φύσης των απειλών. Είναι σχεδόν αδύνατο αν έχουμε επίθεση στον κυβερνοχώρο να διαφοροποιήσουμε αν πρόκειται για στρατιωτική ή μη στρατιωτική επίθεση ή εγκληματική επίθεση. Δηλαδή, αν ε, δείτε ότι χρησιμοποιούνται όλο ένα και πιο πατριωτικές ε, οντότητες ε, από κάποιους ε, και παραδίδουν κάποιες εμπορικές ε, συσκευές στο οργανωμένο έγκλημα. Και Βλέπουμε ότι έτσι γίνονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι ο λόγος που το Κοινοβούλιο πάντοτε ήθελε να διαφοροποιήσει και να διακρίνει το στρατιωτικό από το πολιτικό τμήμα και ακριβώ ε, γι' αυτό το λόγο θέλαμε να έχουμε τη δυτή χρήση. Και το λέω αυτό, γιατί αυτό το πρόβλημα θα το διαπραγματευτούν ε, οι Υπουργοί Έρευνας και η Υπουργή Έρευνα ε, σε διαφοροποίηση από του Υπουργούς Εσωτερικών ήταν πολύ πιο διστακτική. Έτσι λοιπόν, το Κοινοβούλιο θέλει να βρει ένα συμβιβασμό σε τέτοιες πολύπλοκες τροπολογίες δυνάμει της πραγματικότητας και νομίζω ότι θα ήταν ε, κρίμα να χαθούν στο πλαίσιο κάποιων διαπραγματεύσεων γιατί θα είναι περισσότερο οι υπουργοί εσωτερικών που θα διαπραγματευτούν το θέμα αυτό παρά οι υπουργοί έρευνα. Έτσι λοιπόν σα ζητούμε να παρακολουθείτε στενά τη ροή των διαπραγματεύσεων, γιατί οι διαπραγματεύτε μπορεί να μην έχουν μια τέτοια συγκεκριμένη οπτική επί της πραγματικότητα μπορεί να καθοδηγούνται από συστημική διάκριση των τομέων ενώ το Κοινοβούλιο ουσιαστικά είχε προετοιμάσει το δρόμο για ρεαλιστικό συμβιβασμό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, τα σημειώνω. Μάλιστα, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ και πάλι. Θα ήθελα να σας φίξω το χέρι, ήταν πολύ μεγάλη ικανοποίηση που σας είχαμε εδώ. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αγαπητοί φίλοι. Δεν ξέρω Καλά νέα, κακά νέα. Δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντική η απόψη σας για μένα. Ακυρώνεται η αυριανή συνάντηση της Επιτροπής μας. Καλά ή κακά νέα δεν ξέρω. Επομένως, περνάμε στο 19, διάφορα, δεν έχουμε διάφορα, συνεδριά συνεδριάσεις 18 Φεβρουαρίου το απόγευμα και 19 Φεβρουαρίου και το πρωί και το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ και αντίο.